Good Κυρίες και κύριοι, καλώς σας απόγευμα. All Σας ευχαριστώ που ήρθατε εδώ να συζητήσετε μαζί μας σε μια τόσο ηλιόλουστη μέρα. Έχουμε να συζητήσουμε λοιπόν σημαντικά ευρωπαϊκά θέματα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν τη συνεδρίασή μας. Η συνεδρίασή μας ε, θα διαρκέσει μέχρι αύριο το απόγευμα. Θα συνεδριάσουμε αύριο πρωί και απόγευμα. Έκριση τη ημερήσια διάταξη. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, ε, μπορούμε να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Δεν βλέπω να υπάρχουν παρατηρήσει. Σα ευχαριστώ πολύ. Ανακοινώσει του Προέδρου. Ε, ολομέλεια της ενεργειακής κοινότητας. Πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Θα πρέπει να νιώθουμε υπεύθυνοι για την διεθνή συνεργασία εντός της ενεργειακής κοινότητας. Εννέα χώρες από τα Δυτικά Βαλκάνια, η Μολδαβία, η Ουκρανία και η Γεωργία και κάποιοι παρατηρητές θα συμμετάσχουν διότι το 2005 Ήμασταν εμείς ε, η αρμόδια επιτροπή για τη διαδικασία αυτή. Σας καλώ λοιπόν ε, στην Ολομέλεια αύριο ανάμεσα στην πρωινή και απογευματινή μας συνεδρίαση, δηλαδή 24 Απριλίου από τις 1.30 μέχρι τις 2.30. Μία ώρα θα κρατήσει. 1.30 με 2.30. Το APS αίθουσα 3Ε3. Η συνάντηση αυτή ανάμεσα στους βουλευτές της Ήτρε και ε, βουλευτές ε, της ενεργειακής κοινότητας είναι πολύ σημαντική για την συνεργασία μας ε, με τα Δυτικά Βαλκάνια και τις, τους ανατολικούς μας ε, γειτόνους, τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία. Θα ήθελα λοιπόν να σας καλέσω να παρευρεθείτε στην συνεδρίαση αυτή, ακόμα και αν είναι μόνο για μισή ώρα ή για 20 λεπτά. Να έρθετε να ακούσετε τι λέμε. Σας παρακαλώ λοιπόν να είσαστε παρόντες. Ε, θα μιλήσουμε για την ε, βιώσιμη χρήση της ε, ενέργειας στην ενεργειακή κοινότητα. Θα πρέπει να το συζητήσουμε αυτό με τους γειτόνους μας, εάν μας ενδιαφέρει το θέμα αυτό. Ένα σάντουιτς λοιπόν για μεσημεριανό. Θα ευχαριστώ τούν σάντουιτς λοιπόν από τη μία μέχρι τις μία πριν την ε, συνάντηση αυτή. Στην αίθουσα 3ε3 λοιπόν μπορούμε επίσης να φάμε ένα σάντουιτς ε, διότι δεν θα προλάβουμε να φάμε μεσημεριανό αλλού. Σας παρακαλώ λοιπόν να παρευρεθείτε εκεί. ας ε, παραβρίσκονται τουλάχιστον ένας ή δύο ε, συνάδελφοι από τις μεγάλες πολιτικές ομάδες ε, και από ένας από τις μικρές. Κατά την τελευταία τέτοια συνεδρίαση, παρόντες ήταν δύο βουλευτές της Ήτρε, ο Γιάννη και η Ρεμπέκα Χάρμς. Δεν δώσαμε πολύ καλή εικόνα, φανταστείτε. Διότι ήρθαν άνθρωποι ε, από πολύ μακριά, 3.000 χιλιόμετρα, 5.000 χιλιόμετρα για να συναντηθούν μαζί μας και δύο ευρωβουλευτές μόλις ήταν παρόντες. Σας παρακαλώ λοιπόν να παρευρεθείτε έστω και για λίγα λεπτά. Διότι αν θέλουμε να δείξουμε ότι παίρνουμε στα σοβαρά τις δικές μας αποφάσεις, ε, αυτό απαιτείται. Προχωρώ τώρα σε άλλη ανακοίνωση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα οργανώσουν διάσκεψη διαμορφώνοντας ε, το ψηφιακό μας μέλλον, η πρόκληση της ψηφιακή επανάστασης ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες στις 25 Απριλίου από τις 2.30 έω τι 6.30 το απόγευμα. 25 Απριλίου. Τετάρτη. Τετάρτη απόγευμα λοιπόν διαμορφώνοντας το ψηφιακό μας μέλλον η πρόκληση της ψηφιακής επανάστασης. Η διάσκεψη αυτή θα επικεντρωθεί μεταξύ άλλων στις επενδύσεις για να ξεκλειδώσουμε την ψηφιοποίηση και να ε, αποφύγουμε ε, το ψηφιακό χάσμα, την ε, καινοτομία και τις ευκαιρίες για τους Ευρωπαίους πολίτες, καθώς και μια ψηφιακή ενιαία αγορά για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Προσκεκλημένοι είναι όλοι οι ευρωβουλευτές της Ήτρε. Κάποιοι από εσά χαμογελούν ε, ευγενικά. Αυτό δεν το είδα όμως ε, στην ε, πρώτη μου ανακοίνωση. Σας καλώ λοιπόν να συμμετάσχετε και στη συνάντηση για την ενεργειακή κοινότητα και σε αυτήν. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων 21η και 22η Φεβρουαρίου 2018. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσει μέχρι το τέλο τη συνεδρία, θα θεωρηθεί ότι εγκρίνονται τα ε, πρακτικά. Τέταρτο θέμα. Κανονισμός για τον ΕΝΙΣΑ, τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο, δική μας αρμοδιότητα, και την κατάργηση του κανονισμού υπαριθμών 526 του 2013, καθώς και σχετικά με την πιστοποίηση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών. Πράξη για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, με λίγα λόγια. Θα θέλαμε λοιπόν ε, να εξετάσουμε και να εγκρίνουμε το σχέδιο έκθεσης και η συγγήτρια είναι η συνάδελφος Αγγέλικα Νίμπλερ. Έχουμε και εδώ κάποιους σκιώδεις εισηγητές όπως βλέπω. Ωραία. είναι ένα από τα θέματα προτεραιότητας ε, σύμφωνα με την κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Κοινοβουλίου. Η Επιτροπή ε, ε, ΙΜΚΟ ε, είναι συνδεδεμένη Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 54 του κανονισμού με μοιρασμένε αρμοδιότητες στον τίτλο 3 για την πιστοποίηση. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν την συζήτηση. Κυρία Ισηγήτρια, θα σας παρακαλούσα να παρουσιάσετε το σχέδιο έκθεσής σας. Έχετε το λόγο. Κυρία Νίμπλερ. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφοι, χαίρομαι που έχω τη δυνατότητα να σας παρουσιάσω σήμερα ε, την ε, έκθεσή μου για την πράξη για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Θα ε, ήθελα να ευχαριστήσω όσους ήρθαν σε επαφή μαζί μου ήδη πριν την εκπόνηση της έκθεσης αυτής. Σας ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις σας και προσβλέπω στην καλή συζήτηση σήμερα εδώ στην Επιτροπή. Τις τροπολογίες μου θα ήθελα να τις συνοψίσω Τρία θέματα θα ήθελα να αναφέρω. Καταρχάς, τον ρόλο της ΕΝΙΖΑ και την εντολή της. Στο μέλλον πώς θα εργάζεται, τι κατεύθυνση θα έχουν οι εργασίες της. Το δεύτερο θέμα είναι πώς θα τα καταφέρουμε να έχουμε υψηλά επίπεδα κυβερνοασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το τρίτο θέμα που θα ήθελα να αναφέρω είναι πώς θα καταφέρουμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών ε, στις ε, ψηφιακές, ε, τις επιγραμμικές υπηρεσίες. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα για μένα λοιπόν ε, η εμπιστοσύνη των πολιτών. Όσον αφορά την ε, εντολή, ε, από πολιτική άποψη εγώ θα ήθελα μια πιο, έναν πιο ισχυρό ευρωπαϊκό οργανισμό και στηρίζω γι' αυτό την πρόταση της Κομισιόν και όσον αφορά τη χρηματοδότηση και όσον αφορά τον προϋπολογισμό. Επίσης, να δοθεί μόνιμη εντολή στην ΕΝΙΖΑ. Θέλουμε επίσης να ενισχύσουμε το ρόλο της ΕΝΙΖΑ στον έλεγχο και την πιστοποίηση. Και δεν νομίζω ότι αυτό ε, αντίκειται στον ισχυρό ρόλο που έχει να παίξει για την κυβερνοασφάλεια. Ε, στην Ευρώπη κάποιοι εθνικοί οργανισμοί εργάζονται πολύ καλά, σε άλλες χώρες όμως αυτή τη στιγμή δημιουργούνται οργανισμοί κύβερνο ε, με βάση την ε, ε, οδηγία για την ασφάλεια στο ε, διαδίκτυο που εγκρίναμε πριν κάποιο καιρό εδώ. Θέλουμε λοιπόν πιο, ισχυρή, πιο ισχυρό οργανισμό, πιο ισχυρή εντολή και θέλουμε επίσης να ενθαρρύνουμε τη συνεργασία ανάμεσα στην ΕΝΗΣΑ και τους εθνικούς οργανισμούς και έχω υποβάλει σχετικές προτάσεις. Πιστεύουμε λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρχει ισχυρή επιχειρησιακή συνεργασία. Ε, θα πρέπει να οικοδομήσει, να δημιουργήσει επιρρογνωσία η ε, ενίσα και να βοηθήσει και τα κράτη-μέλη σε αυτό. Και επίσης ε, θα πρέπει να δημιουργηθούν ε, ευρωπαϊκά προγράμματα κυβερνοασφάλειας σε συνεργασία με τους εθνικούς οργανισμούς και με άλλους ενδιαφερομένους. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τον ρόλο της ΕΝΙΣΑ. Κύριε Πρόεδρε, μου απομένουν κάποια λεπτά ακόμα. Προχωράω στο δεύτερο θέμα. Πώς θα διασφαλίσουμε υψηλά πρότυπα κυβερνοασφάλειας τι έχω τροποποιήσει στην πρόταση της Κομισιόν. Καταρχάς, ε, έχω τροποποιήσει το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Δεν θα πρέπει να καλύπτονται μόνο οι υπηρεσίες και τα προϊόντα, αλλά το συνολικό ε, ψηφιακό οικοσύστημα και οι διαδικασίες θα πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής. Ελπίζω ε, οι συνάδελφοι να μπορούν να στηρίξουν τον ορισμό που έχω δώσει. Δεύτερον, ε, θέλω μία προσέγγιση που να βασίζεται στον κίνδυνο, όχι ένα μέγεθος για όλους. Θα πρέπει να καθορίσουμε λοιπόν ε, τα επίπεδα ασφαλείας. Κάτι που αντικατοπτρίζεται και στα προγράμματα. Και έχω διατηρήσει την πρόταση της Κομισιόν που βρίσκω καλή όσον αφορά τα τρία επίπεδα ασφαλείας που προτείνει. Προσπάθησα να διατυπώσω ε, με μεγαλύτερη σαφήνεια τα επίπεδα ασφαλείας αυτά και θα ήθελα πολύ να ακούσω τις παρατηρήσεις των συναδέλφων, αν και εκείνοι συμφωνούν ή θεωρούν ότι θα πρέπει να γίνουν περαιτέρω προσαρμογές. Και φτάνω στο θέμα της πιστοποίησης. Αυτό πώς θα το διαμορφώσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό ήταν δύσκολο θέμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήθελε ε, θελούσια προσέγγιση σε όλο το φάσμα. Εγώ ε, έχω επιλέξει την μέση οδό, ακριβώς αυτή την προσέγγιση που βασίζεται στον κίνδυνο, την οποία θεωρώ καλύτερη. Και εδώ θα με ενδιαφέρε να ακούσω τη γνώμη των συναδέλφων. Πάντα μιλάμε για τις συνδεδεμένες συσκευές, ε, τις ε, συσκευές που είναι συνδεδεμένες με το διαδίκτυο, όπου υπάρχει υψηλός κίνδυνος. Εδώ λοιπόν ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε ένα υποχρεωτικό σύστημα για τα άλλα δύο ε, επίπεδα να είναι προαιρετικό και μάλιστα στο χαμηλότερο επίπεδο ασφαλείας ε, να υπάρχει και η δυνατότητα αυτοπιστοποίησης. Αυτή λοιπόν είναι η δική μου πρόταση. Είναι όμως πολύ επίμαχο το θέμα και υπάρχουν πολλές διαφορετικές απόψεις. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω την απόψη των συναδέρφων. Από τη μία θέλουμε υψηλό επίπεδο ασφαλείας και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικό σύστημα πιστοποίησης. Διότι αλλιώς μπορεί να μην έχει και κίνητρο για πιστοποίηση. Από την άλλη όμως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν θα πρέπει να δημιουργήσουμε εμπόδια εισόδου στην αγορά. Μιλάμε για εκατομμύρια συσκευέ ε, που θα μπορούσαν να εμπίπτουν εδώ και ε, εάν είναι υποχρεωτική η πιστοποίηση. Πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, μπορούν να θεωρήσουν ότι διαρκεί υπερβολικά η διαδικασία της πιστοποίησης. Γι' αυτό εγώ προτείνω τον συγκεκριμένο συμβιβασμό. εξέτασα και το άρθρο 49, όπου ρυθμίζεται η σχέση του ευρωπαϊκού με τα εθνικά συστήματα. Η Κομισιόν προτείνει να αντικατασταθούν τα εθνικά συστήματα από το ευρωπαϊκό. όσον αφορά τη σχέση των εθνικών οργανισμών με τον ε, ΕΝΙΖΑ έχω υποβάλει σχετικές ε, τροπολογίες ε, και το τελευταίο θέμα είναι πώς θα πετύχουμε τη συμμετοχή και των κρατών μελών ε, και των βιομηχανιών στη διαδικασία επιστοποίησης. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, έχει συζητηθεί ιδιαίτερα η συμμετοχή των stakeholders των ενδιαφερομένων της βιομηχανίας. εκατοντάδες ε, εργαζομένους ε, αφορά το θέμα αυτό. Εμείς αυτή τη στιγμή έχει 60 με 80 άτομα προσωπικό. Ε, εάν λάβουμε υπόψη και τους συνεργαζόμενους φορείς, μιλάμε για εκατοντάδες. Χωρίς συμμετοχή των ενδιαφερομένων δεν θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ικανοποιητικά επίπεδα ασφαλείας. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε πώς μπορούμε με έξυπνο τρόπο να πετύχουμε την συμμετοχή ε, των βιομηχανιών, των ενδιαφερομένων. Ο πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια. Προτείνω λοιπόν ε, ένα πλαίσιο όπου να μπορούν ε, να υποβάλουν τις απόψεις τους τα κράτη-μέλη και επίσης συμμετοχή ad hoc πλατφόρμας ε, για τις ε, βιομηχανίες. Και επίσης όσον αφορά την εμπιστοσύνη των πολιτών ε, δεν προτείνω εδώ συγκεκριμένη επισήμανση αλλά υποχρεωτική δήλωση προϊόντος. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ελπίζω να έχουμε μια ενδιαφέρουσα ανοιχτή συζήτηση από το SND ο έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω καταρχήν που μας υπενθυμίσατε αυτήν την εκδήλωση όπου η Μολδαβία και άλλες χώρες των Βαλκανίων θα συμμετάσχουν. Ξέρετε ότι αποτελεί προτεραιότητα της Βουλγαρικής Προεδρίας εμείς στην Ανατολική Ευρώπη γνωρίζουμε πολύ καλά πόσο σημαντικό είναι να συμμετέχουμε σε τέτοιες συνεδριάσεις. Θα ήθελα λοιπόν να, να συγχαρώ την κυρία Νίμπλερ. Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Γνωρίζουμε ότι η Γερμανία θέλει μια πιο ισχυρή, μια καλύτερη ενίσα και η κυρία Νίμπλερ ε, έχει την ίδια θέση. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, είναι πολύ σοβαρή. Υπάρχει μια πρόταση αύξηση του προπολογισμού από τα 11 στα 23 εκατομμύρια. Νομίζω θα χρειαστούμε βεβαίως και άλλα χρήματα. Θα πρέπει οπωσδήποτε να ενισχύσουμε το ρόλο της ΕΝΗΣΑ ε, προς τρεις κατευθύνσεις. Πρώτα απ' όλα η ΕΝΗΣΑ πρέπει να μπορεί να αναλύσει τις διάφορες απειλές και τις διάφορες ε, πηγές πληροφοριών, περισσότερο εξοπλισμό, τεχνικό εξοπλισμό ε, και επίσης η ΕΝΗΣΑ θα πρέπει να συντονίζεται καλύτερα με τους άλλους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να είναι υπεύθυνη η ενίσα για το blueprint, δηλαδή να δημιουργήσει ένα πλαίσιο εντός του οποίου θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις επιθέσεις από διάφορες, ε, διάφορων τύπων επιθέσεων, επιθέσεις τέλο πάντων, από διάφορες πηγές. Ε, καθώς δημιουργείται αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει η ΕΝΙΣΑ να έχει τη δυνατότητα να αντιδράσει απέναντι σε επιθέσεις ε, που δέχονται διάφορα κράτη-μέλη και ο διευθυντής πρέπει να λογοδοτεί. Πρέπει να λογοδοτεί στο Κοινοβούλιο και θα πρέπει να είναι και ειδικό σύμβουλος ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε χώρες όπως η Γαλλία ή η Σιγκαπούρη, ο επικεφαλής της ε, υπηρεσίας κυβερνοασφάλειας είναι και άμεσα υπεύθυνος, ε, έχει άμεση επαφή με τον Πρωθυπουργό της χώρας. Πρέπει η Ενίσα να μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε τον εγωισμό κάποιων κρατών μελών. Σε ό,τι αφορά τώρα τη διαδικασία πιστοποίησης, εγώ θα έλεγα να δημιουργηθεί μια νέα ομάδα εργασίας. Θα πρέπει να υπάρχει μια ομάδα ε, στην οποία θα συμμετέχουν διάφοροι εμπλεκόμενοι φορείς, ε, εκπρόσωποι των επιχειρήσεων παραδείγματο χάρη, θα πρέπει να υπάρχουν προγράμματα θελοντικής πιστοποίησης και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με το πώς ορίζουμε τις διάφορες έννοιες, διότι ορισμένε φορές η κυβερνοασφάλεια μπορεί να οδηγήσει σε φόβους. Θα ήθελα να συμφωνήσω με του αδέρφου ε, της Επιτροπής ΙΜΚΟ και την πρότασή τους. Οι διάφορες μονάδες πιστοποίησης θα πρέπει να παρακολουθούν ε, άλλες μονάδες πιστοποίησης που είναι πιο αδύναμες και να τις βοηθούν. Και η ενίσα πρέπει να μπορεί να υποπτεύει τις πιο αδύναμες αυτές ε, υπηρεσίες ε, και εκεί όπου δεν υπάρχουν να βοηθήσει στη δημιουργία, τη δημιουργία τους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ συνάδελφε για τα σχόλια. Ο επόμενος ομιλητής ε, είναι ο κ. Εύγεν Τοσανόφσκι, η Ευγέν Τοσανόφσκι από την ECR. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας πω ότι εκτιμώ την έκθεση της κυρίας Νίμπλερ. Ε, είναι μια πολύ καλή βάση για τις εργασίες στην Επιτροπή μας. Υποστηρίζω και προ, τις προτάσεις βελτίωσης που η ίδια έχει υποβάλει στην έκθεσή της θα πρέπει η ΕΝΙΣΑ να έχει μία μόνιμη εντολή να ενισχυθεί σε επίπεδο ανθρώπινων αλλά και οικονομικών πόρων διότι ο κόσμος στον οποίο ζούμε είναι όλο και πιο περίπλοκος και τα πεδία μάχης ε, δεν είναι αυτά που ήταν στο παρελθόν οι μάχες δίνονται συχνά πλέον ε, σε ένα ψηφιακό περιβάλλον και είναι δύσκολο κανείς ε, να οργανωθεί σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Ε, χαίρομαι επίσης που γίνεται αναφορά στο σύστημα πιστοποίησης των διαδικασιών. Τώρα υπάρχουν κάποια σημεία που δημιουργούν ερωτηματικά, αλλά αυτά μπορούν να συζητηθούν σε επίπεδο σκιωδών φυγητών ο ρόλος συντονισμού και υποστήριξης της ΕΝΗΣΑ είναι σαφής αλλά έχω και ένα ερωτηματικό σε ό,τι αφορά τις επιχειρησιακές ε, λειτουργίες, τις επιχειρησιακές ε, ε, δυνατότητες, διότι θα είναι δύσκολο θα, και θα είναι περίπλοκο αν δώσουμε μια τέτοια αρμοδιότητα στην ΕΝΗΣΑ. διότι θα πάει κάποιος σε, ένα, μια εθνική υπηρεσία να αρχίσει να διατάσει εκεί ε, θα πρέπει να το προσέξουμε αυτό να σκεφτούμε ποιος θα είναι ο αντίκτυπος διότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει έτσι, επιφυλάξεις στα κράτη-μέλη. Επίσης, ό,τι αφορά την διασυνοριακή κρίσιμη υποδομή, τις χρήσιμες υποδομές και τους σχετικούς ελέγχους αυτό είναι ένα δύσκολο ζήτημα το οποίο θα μας ε, ε, οδηγήσει σε περίπλοκες συζητήσεις. Η ΕΝΙΣΑ βεβαίως είναι ε, υπεύθυνη για το συντονισμό των εθνικών συστημάτων εκπαίδευσης στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, κατάτησης δηλαδή. Βεβαίως υπάρχει ανισορροπία μεταξύ των διαφορών χωρών. Κάποιες χώρες είναι πολύ πιο προχωρημένες από άλλες θα πρέπει να υπάρξει μια εξισορρόπηση σε ό,τι αφορά τώρα την πιστοποίηση για αυτό που είπε η συγγήτρια. Εμείς ε, υποστηρίζουμε μια εθελοντική προσέγγιση. Αντιλαμβάνομαι την πρόταση της συγγήτριας να βασιστούμε στο κίνδυνο, στην αξιολόγηση του κινδύνου, αλλά ίσως να πρέπει να το αντιστρέψουμε αυτό. Η αξιολόγηση του κινδύνου ορισμένε φορές υποτιμάται ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε επίπεδο Ένωση. Ένωσης. Ε, και πολλά ζητήματα δεν βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα, σε επιστημονική αξιολόγηση των δεδομένων ε, όπως στις ΗΠΑ παραδείγματος χάρη οι Αμερικανοί βασίζονται σε μια αξιολόγηση του κινδύνου και όταν αξιολόγηση δείχνει ότι μια υποδομή απειλείται τότε περνάμε σε ένα υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας. Εμείς μάλλον αυτήν την προσέγγιση προτιμούμε. Συμφωνούμε με τη δημιουργία των, της πλατφόρμας α, διαβούλευσης ε, στο 47 είναι αυτά, αλλά δεν ξέρω πού θα μπορούσε να εισαχθεί αυτό. Υπάρχει ε, η ομάδα με τα μόνιμα μέλη, υπάρχει δική μας ομάδα, πρέπει να δούμε πού θα τοποθετηθεί αυτή η πλατφόρμα. Και τέλος, θα πρέπει να υπάρξει μια εξισορρόπηση των διαφόρων επίπεδων ασφαλείας. Νομίζω ότι ε, δεν πρέπει να είμαστε υπερβολικά λεπτομερείς στην περιγραφή μας, διότι τα πράγματα αλλάζουν γρήγορα. Ε, έχουμε εξελίξεις σε αυτό το τομέα και πρέπει να παραμείνουμε ευέλικτοι ευέλικτη και στο μέλλον με βάση τις εμπειρίες που θα αποκομίσουμε ενδεχομένως να μπορέσουμε να οδηγηθούμε σε, μια έναν οριζόντιο ορισμό. Θα πρέπει επίσης να εγγυηθούμε ότι θα υπάρχει μια συνέπεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό έχει να κάνει με ένα σύστημα το οποίο αυτή τη στιγμή δεν είναι ισορροπημένο και συμφωνώ με την εισηγήτρια ότι αυτή η διαδικασία θα πρέπει να οριστεί σαφώς. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά την εισηγήτρια, γιατί είναι μια εξαιρετικά ποιοτική ε, έκθεση αυτή που μας παρουσίασε. Ευχαριστώ πολύ. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κ. Παύλ Τέλιτσκα από τους φιλελεύθερους στην άλλη, παρακαλώ. Thank you, Chair. Uh, Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Νίμπλερ. Στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων δεν θέλω να αναφέρω όλα τα σχολιά μου, απλώς θα επικεντρωθώ σε κάποια σημεία και στη συνέχεια σε άλλες συναντήσεις των σχεδόν. Θα έχουμε την ευκαιρία να σχολιάσουμε λεπτομερέστερα και σε κάποιο βαθμό θα εισαγάγουμε και τις τροπολογίες που θα αναφέρω. Κάποιες παρατηρήσεις τώρα σε ό,τι αφορά το ρόλο του ΕΝΙΣΑ. Νομίζω ότι η κατεύθυνση που ακολουθεί η συγγετρία είναι μια πολύ λογική κατεύθυνση, η γραμμή που ακολουθεί. Νομίζω ότι η πλειοψηφία ημών θα συμφωνήσει ότι δεν επιζητούμε πλήρη επανάσταση, αλλά θέλουμε έναν ισχυρό, σταθερό μόνιμο οργανισμό που να είναι καλά εξοπλισμένος. Η ερώτηση που θα θέσω είναι μήπως ε, θα πρέπει να προσπαθήσουμε στην έκθεση αυτή να μην ε, υπογραμμίσουμε τη μελλοντική εξέλιξη του ΕΝΙΣΑ γιατί όλο το οικοσύστημα του, ε, του κυβερνοχώρου θα αλλάξει και δεν μπορούμε να προβλέψουμε σήμερα τι θα χρειαστεί σε ένα-δύο χρόνια. Ίσως ε, να πρέπει να έχουμε και μία ρήτρα αναθεώρηση ε, που θα λέει σε τι θα πρέπει να επικεντρώνεται η επόμενη αναθεώρηση. Και ε, νομίζω ότι σε κάποιες εκτιολογικές σχέσεις θα μπορούσαμε να έχουμε ένα τέτοιο σύνδεσμο. Η φιλοδοξία μας λοιπόν είναι να το έχουμε αυτό υπό έλεγχο και να έχουμε εσωτερική δυναμική για το μέλλον. Δεύτερη παρατήρηση. Σε ό,τι αφορά το ρόλο, κατά τα λοιπά, Νομίζω ότι με όσα προτάθηκαν θα συμφωνήσουμε σε γενικές γραμμές. Τώρα, άλλα σχόλια για το επίπεδο της ασφάλειας. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το δούμε εις βάθος, έτσι ώστε να κατανοούμε ένας τον άλλον. Γιατί, από ό,τι καταλαβαίνω, η εισηγήτρια προτείνει υψηλή ασφάλεια. Εγώ θεωρώ ότι ήδη φύγουμε το θέμα της εθνικής ασφάλειας που είναι πέραν του πεδίου εφαρμογή ε, αυτού του σχεδίου νομοθεσίας. Όμως ε, οι διαβουλεύσεις μεταξύ των σκιωδών ε, θα μας δείξουν τι σκέφτεται ακριβώς η συγγήτρια για το θέμα αυτό. Χαίρομαι που η συγγήτρια αναφέρθηκε στο θέμα της δομής του θεσμού ακόμη και αν μπορεί να χρειαστεί να υπάρξει κάποια προσέγγιση των θεσεών μας. Όμως ε, είναι καλό που πιστεύει ότι η δέσμευση των κρατών μελών, ε, των οργανισμών του, των stakeholder και των καταναλωτών πρέπει να υπάρχει και όλοι ξέρουμε ότι όλοι θα θέλουν να συμμετέχουν, όμως θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε μία δομή που να λειτουργεί. Και επίσης θα πρέπει να σκεφτούμε το ποιος θα έχει και ποιο ρόλο. Δηλαδή να προσδιορίσουμε την ανάγκη των συστημάτων, των προγραμμάτων. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε λίγο παραπέρα από αυτό που προτείνει η Κομισιόν, γιατί ε, θα ήμουν ε, πολύ διστακτικός ε, στο να δημιουργήσουμε διάφορες δομές, όμως ο κλάδος ξέρει πολύ καλά ποιες είναι οι ανάγκες. Χρειαζόμαστε λοιπόν αλληλεπίδραση για να βρούμε συγκεκριμένες λύσεις και ευχαρίστως να προτείνω κάτι προς αυτή την κατεύθυνση. Το θέμα της απόρριψης θέτει κάποιες δυσκολίες σε μένα, όμως θα διερευνήσουμε καλύτερα το ποια κατεύθυνση μπορούμε να ακολουθήσουμε. Σε ό,τι αφορά τη δήλωση προϊόντος, αυτό είναι ένα ακόμα ανοιχτό θέμα που θα πρέπει να εξετάσουμε. Χαίρομαι και πάλι που η εισηγήτρια έδειξε το θέμα. Όμως, ίσως ε, να έχω κάποιες προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Και τώρα, τελευταία παρατήρηση. Μία από τις ε, μεγαλύτερες δυσκολίες θα είχα σε σχέση με το εκούσιο σύστημα τι ακριβώς εννοείται πρέπει να καταλάβω. Όμως η κυρία Νίμπλερ είπε ότι πρόκειται για ένα υβριδικό σύστημα αυτό που προτείνει. Αυτό μέσα σε εισαγωγικά. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Θα πρέπει να έχουμε είτε ένα ακούσιο σύστημα είτε ένα υποχρεωτικό σύστημα και ίσως θα πρέπει να διαλέξουμε το θελοντικό αλλά με εσωτερική δυναμική για το μέλλον. Δηλαδή να μπορεί να υπάρξει δυνατότητα τροποποίησης. Τελειώνω, Πρόεδρε γιατί νομίζω ότι θα έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε και θα παρουσιάσω κάποιες τροπολογίες. Όμως ε, είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσουμε να έχουμε προσέγγιση των θεσεών μας ε, και ανυπομονώ γι' αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ για το καλό σχέδιο κειμένου. Ευχαριστούμε για την ομιλία σας. Πάμε λοιπόν τώρα στους λοιπούς ομιλητές, ομιλητές. Ευχαριστώ, Αγγέλικα, για την εξαιρετική έκθεση. Δεν είναι κάτι εύκολο, αλλά είναι ισορροπημένο το κείμενο. Θα πρέπει να σκεφτούμε πώς ε, θα προσανατολιστούμε καλύτερα απέναντι σε κάποιες λύσεις. Καταρχήν, συμφωνώ ότι η ΕΝΙΣΑ θα μπορούσε να παίξει ρόλο κλειδί στο να προωθήσει την ασφάλεια στον κυβερνό χώρο και να υπάρχει καλύτερη σχέση μεταξύ των διάφορων και δημόσιων ενδιαφερομένων μερών. Θα πρέπει λοιπόν να το τονίσουμε αυτό. Από την άλλη όμως νομίζω ότι θα πρέπει να καταστήσουμε πιο σαφή το ρόλο της ΕΝΙΣΑ σε ό,τι αφορά την υιοθέτηση του συστήματος πιστοποίησης, του προγράμματος πιστοποίησης και για το ε, ε θα προτείνει το αν υπάρχει ανάγκη για ε, την ύπαρξη τέτοιων συστημάτων πιστοποίησης. Θα πρέπει λοιπόν να έχει ένα ζωτικό ρόλο η ΕΝΙΣΑ σε αυτό το θέμα. Δεύτερον, Πιστεύω ότι έτσι όπως ε, προτάθηκε από την Κομισιόν και όπως ε, έχουμε στην έκθεση, όπως προτείνεται από την Αγγελικά, θα πρέπει να υποστηρίξουμε και τον κλάδο στη διαδικασία της πιστοποίησης θα πρέπει να είναι πολύ πιο σαφές από την έποψή μου ότι η μόνιμη ομάδα των ενδιαφερομένων ε, θα πρέπει να συζητήσει με ε, τους παρόχους ε, και ίσως θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε και τους καταναλωτές, να είναι πιο ευρύ αν θέλουμε να έχουμε και κάποια ομάδα συμβουλευτική. Επίσης, πιστεύω ότι η μόνιμη ομάδα των ενδιαφερομένων μερών ε, θα πρέπει να έχει την ε, αρμοδιότητα να προτείνει συστήματα πιστοποίησης και να διαβουλεύεται την ενίσα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προορισμού των συστημάτων αυτών. Νομίζω ότι θα ήμασταν πιο κοντά στο να κατανοήσουμε ότι δεν υπάρχει μια λύση που να ταιριάζει σε όλους. Πρέπει να εργαστούμε ανά περίπτωση και να βασιζόμαστε στα επιτεύγματα του κλάδου. Χρειαζόμαστε φυσικά πιστοποίηση και σε κατώτερο επίπεδο. Είναι σαφές όταν συμφωνούμε για το υψηλότερο επίπεδο θα πρέπει να σκεφτούμε τι θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό αλλά από την άλλη είμαι κάπως ε, προσεκτικός, γιατί υπάρχουν πολλές απαιτήσει. Όμως, σε μια τελογική σκέψη θα ήθελα να περιλαμβάνεται ο χάρτης πορείας προς τις υποχρεωτικές λύσεις. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μούλτη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την εισηγήτρια και τους σκιώδεις εισηγητές. Ανέφεραν πολλά σημαντικά σημεία στην έκθεση αυτή. Ένα παράδειγμα είναι οι τροπολογίες στην πρόταση της Κομισιόν που αναφέρονται στην ασφάλεια εξχεδιασμού. Κάτι που είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Γιατί δεν μιλάμε μόνο για το τελικό προϊόν και τις υπηρεσίες που θα πρέπει να πιστοποιηθούν, αλλά και ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη είναι ζωτικά σε αυτό το έργο. Ένα άλλο θέμα ανησυχίας αφορά το κόστος ε, της αξιολόγησης και της πιστοποίησης για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει. Πριν το χάρη, αν δούμε ένα είδος αυτοαξιολόγησης για τις ΜΜΕ στη διαδικασία αυτή. Ένα άλλο θέμα αφορά τη φύση και το εύρος της κυβερνοασφάλειας. Τι σημαίνει δηλαδή αυτό θα μπορούσε να αφορά και μεμονωμένα νοικοκυριά ή κρίσιμες υποδομές. Επίσης, ε, τονίστε και η ανάγκη να υπάρχει συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, όπως το ΝΑΤΟ, προηγούμενος χάρη, και ο σκοπός της πιστοποίησης είναι να αυξηθεί η εμπιστοσύνη, κάτι που είναι ευκταίο. Όμως υπάρχει και ένας ενδυνάμει κίνδυνος η πιστοποίηση να οδηγήσει σε ανοχή. Δεν θέλουμε οι καταναλωτές να πιστεύουν ε, ότι ότι είναι ασφαλείς καταναλωτές επειδή θα έχει μια υψηλή βαθμολόγηση το προϊόν και θα υπάρχουν κάποια τροτά σημεία που θα εμφανιστούν κατόπιν της διαδικασίας πιστοποίησης. Παραδείγματο χάρη, αν δούμε τους κινδύνους ε, της, ε, των συνδέσεων που μπορεί να οδηγήσουν σε μετέπειτα τροτά σημεία. Ε, οι τροπολογίες, έχουν κατατεθεί κάποιες τροπολογίες για να καθορίσουν τη σημασία ε, ουσιαστικά του αλφαβητισμού ε, στον κυβερνοχώρο. Δεν είχα λοιπόν πολλά προσθέσω. Πολύ καλή δουλειά. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής, η κυρία Γκροστέ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να συγχαρώ την εισηγήτρια την Αγγέλικα που έκανε μια πολύ καλή δουλειά για ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα πρέπει όντως να ενισχύσουμε οπωσδήποτε τον ρόλο της ΕΝΙΣΑ έτσι ώστε να γίνει μια πραγματική ευρωπαϊκή υπηρεσία που να είναι σημείο αναφορά στον τομέα τη κυβερνοασφάλεια. Πρέπει λοιπόν να ενισχυθεί η πραγματογνωμοσύνη τη για μια καλύτερη προστασία απέναντι στι κυβερνοεπιθέσει. Ε, θα πρέπει επίση να παίζει ένα ρόλο, ε, ένα σαφή ρόλο ευαισθητοποίηση για τα συγκεκριμένα αυτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην κοινή γνώμη, η προηγούμενη εντολή τη ΕΝΗΣΑ ήταν ε, εξαιρετικά ασαφή. Είναι λοιπόν η ευκαιρία όλα αυτά να διευκρινιστούν. Μίλησαν όλοι για, τις, για το επίπεδο πιστοποίηση. Ε. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να είναι προσαρμοσμένο αυτό το επίπεδο, διότι οι κίνδυνοι δεν είναι οι ίδιοι ανάλογα με τον κάθε τομέα και με το κάθε προϊόν. Η υποχρεωτική πιστοποίηση, η γενικευμένη, ε, αυτόματη, σίγουρα θα δημιουργήσει σημαντικό διοικητικό άχθος το να συνδέσουμε όμως ένα ηλεκτρονικό δίκτυο ή ένα αεροδρόμιο ε, δεν είναι το ίδιο, είναι άλλες οι ανάγκες. Ε, ε, εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να έχουμε διάφορα επίπεδα ασφάλειας ανάλογα με τον κίνδυνο και, να, βεβαίως να ορίζονται σαφώς αυτοί οι κίνδυνοι. Σε ό,τι αφορά το επίπεδο προστασίας, εγώ θα ήθελα να, προστα... να... να προσθέσουμε και κάποια τεστ αποτελεσματικότητα για να μπορούμε να δοκιμάσουμε την ανθεκτικότητα. Είτε μιλάμε για ένα προϊόν, για μια υπηρεσία, για μια διαδικασία. Ανθεκτικότητα απέναντι σε περίπλοκε, προχωρημένε επιθέσει, διότι αν δεν γίνουν αυτά τα τεστ ανθεκτικότητα θα είναι δύσκολο να γνωρίζουμε και πόσο ευάλωτο είναι το σύστημα. Τελειώνοντα, να πω ότι πρέπει ούτω ή άλλω να αποφύγουμε οποιαδήποτε εξίσωση προ τα κάτω σε ό,τι αφορά την ε, κυβερνοασφάλεια πρέπει να επιτρέψουμε στα κράτη-μέλη να πάνε πιο πέρα, πιο μακριά, να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη που έχουν μείνει πίσω ε, να φτάσουν στο επίπεδο των υπολείπων. Συγχαρητήρια πάντω στην εισηγήτρια. Uh, Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Λόπες Περμέχο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η συνάδελφος Μαρίσα Ματίας ε, δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα το απόγευμα, έτσι λοιπόν θα παρέμβω εγώ ε, στο όνομά της, ε, για λογαριασμό της. Σε ό,τι αφορά τώρα την ενίσα, εμείς υποστηρίζουμε την ενίσχυση της επιχειρησιακής δυνατότητας της υπηρεσίας αυτής, της οποίας η εντολή πρέπει να γίνει σεβαστή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε ό,τι έχει να κάνει με την κυβερνοασφάλεια. Θα πρέπει να μπορούμε να απαντήσουμε γρήγορα και συντονισμένα απέναντι σε ενδεχόμενες κυβερνοεπιθέσεις που θα μπορούσαν να λάβουν χώρα στον ευρωπαϊκό χώρο. Και γι' αυτό η ΕΝΗΣΑ πρέπει να υποστηρίξει τα κράτη-μέλη, να του δώσει τη δυνατότητα να απαντήσουν σε τέτοιου είδου επιθέσεις. Βεβαίως η δυνατότητα ε, η αρμοδιότητα για τι αποφάσει πρέπει να παραμείνει σε επίπεδο κρατών μελών. Πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα ε, τον δρόμο που θα ακολουθήσουμε, να μην πέσουμε δηλαδή ε, τον πειρασμό στρατηγικών ε, εποπτείας και παρακολούθησης που να διακυβεύει το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι ένα κοινό ε, αγαθό η ασφάλεια, δεν πρέπει η πολιτική του φόβου να χρησιμοποιηθεί κατά των πολιτών και της ιδιωτικής ζωής. ό,τι αφορά την ε, κυβερνοασφάλεια, εμείς θέλουμε να υπάρχει ένα τέτοιο σύστημα ε, για να γνωρίζουμε ε, ποια προϊόντα είναι ασφαλή και ποια όχι σε επίπεδο κυβερνοασφάλεια. Ιδιαίτερα όταν μιλάμε για προϊόντα τα οποία ε, απευθύνουν, οι υπηρεσίε που απευθύνονται προ του ανήλικου. Πρέπει όμω να συνεργαστεί ενίσα με όλα τα μέσα τα οποία ε, εμπλέκονται στην παραγωγή και την κατανάλωση αυτών των προϊόντων και όχι σε, μόνο σε αυτού που ανήκουν ε, στι μεγάλε επιχειρήσει. Οργανώσει καταναλωτών, μη κυβερνητικέ οργανώσει, μικρομεσαίε επιχειρήσει πρέπει να συμμετάσχουν σε διαφανεί, δημόσιε ε, και συμπεριληπτικέ διαδικασίε. Εμεί θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα μοντέλο πιστοποίηση υποχρεωτικό, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα προϊόντα μέσου και υψηλού κινδύνου. Όλα τα προϊόντα πρέπει να μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλειά του. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο, ένα ελάχιστο πλαίσιο προποθέσεων που θα πρέπει να πληρούν όλα τα προϊόντα για να μπορούν να ρεθούν σε εμπορία στον ευρωπαϊκό χώρο. Αυτό λοιπόν που προέχει εδώ είναι η προστασία των χρηστών που είναι αυτή τι που θα χρησιμοποιήσουν το προϊόν και προ αυτή την κατεύθυνση θα υποβάλουμε και τι όποιε τροπολογίες. Ευχαριστώ. Thank you. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτή ήταν λοιπόν η επίσημη θέση της ΚΟΕ. Σας ευχαριστώ. Και προχωράμε στον επόμενο ομιλητή, τον κύριο Εντουάρτ Μαρτά. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και την εισηγήτρια για το έργο της. Δεν θα επαναλάβω όσα είπαν οι συνάδελφοι. Απλώς θέλω να φερθώ σε δύο σημεία που θεωρώ σημαντικά. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε στο ποιο είναι το τίμημα ε, που θέλουμε να θέσουμε για μια αυξημένη ασφάλεια. Υπάρχουν φυσικά πολλά επίπεδα. Με εκπλήσει η πρόταση Κομισιόν που λέει επίπεδο 2 ε, επίπεδο 2 καλύτερο από το 1, το 3 καλύτερο από το 2 κτλ. Αυτό δεν μας εξηγεί και πολλά. Ευτυχώ ε, που πηγαίνουμε προς τα πάνω, αλλά θα ήθελα ε, να έχουμε κάποιες επεξηγήσεις και τεχνικό προσανατολισμό. Όλα αυτά δεν είναι σαφή. Εγώ τι θα ήθελα και το λέω από την αρχή ότι θα πρέπει να σκοπεύσουμε στο καλύτερο επίπεδο ασφάλειας. Έχουμε χώρες που τα έχουν καταφέρει πολύ καλά. Επίσης, ε, δεν θα πρέπει να βάλουμε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο παντού και συνεχώς, εντάξει, συμφωνώ, όμως και θα πρέπει να έχουμε στο υψηλότερο επίπεδο και νομίζω ότι είπε η κυρία Γκροστέτ, θα πρέπει να έχουμε ένα σύστημα πιστοποίησης που να ανταποκρίνεται σε πραγματικές ε, ανάγκες για να είμαστε σίγουροι ότι το επίπεδο αυτό δεν θα μπορεί να καταστρατηγηθεί. Κατόπιν, αυτό που προτείνει η συγγήτρια, ότι σε ένα μικρότερο επίπεδο μπορούμε να είμαστε λιγότερο και να έχουμε αυτοπιστοποίηση. Εδώ έχω ε, κάποια αμφιβολία γιατί η ε, διαδικασία αυτή της αυτοπιστοποίησης ε, θα καθησυχάσει τον πελάτη. Το αμφιβάλλω επίσης μπορεί να έχουμε πιο εύθραστο επίπεδο ασφάλειας για τις ΜΜΕ. Έτσι λοιπόν μπορεί να κοστίσει παραπάνω. Ποιο είναι λοιπόν το τίμημα που θέλουμε να θέσουμε το θέμα της κυβερνοασφάλειας και αν στοχεύσουμε σε μια κυβερνοασφάλεια low cost, να ξέρετε, οι Κινέζοι θα είναι πολύ πιο ανταγωνιστικοί από εμά. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κούμπουλα Νάτρη. Σας ευχαριστώ πολύ. Η συγγήτρια έχει εργαστεί πολύ πάνω στο θέμα αυτό. Θα ήθελα να θίξω κάποια θέματα. Ε, ξεκινήσαμε το θέμα αυτό όταν βρισκόμασταν στη φάση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και είχαμε πει τότε ότι χρειαζόμαστε ε, τομέα βιοασφάλειας, κυβερνοασφάλειας ε, στην Ευρώπη και θα πρέπει να φροντίσουμε να μην κάνουμε διαφορετικά πράγματα το κάθε κράτος μέλος. Γι' αυτό χρειάζεται συντονισμός. Ταυτόχρονα θα πρέπει να βρούμε τους τεχνικούς τρόπους να το πετύχουμε αυτό. Ε, χρειαζόμαστε καινοτομία διότι ε, και οι εγκληματίες ε, συνέχεια προχωράνε. Πρέπει λοιπόν και εμείς να βρούμε τα ανάλογα μέσα για να τους αντιμετωπίσουμε. Κάθε επιχείρηση που ασχολείται με τα προϊόντα αυτά θα πρέπει να, γνωρίζετε, να γνωρίζει ότι χρειάζονται ε, νέε πληροφορίε και για τους καταναλωτές. Ε, χρειαζόμαστε λοιπόν προσέγγιση που να βασίζεται στον κίνδυνο. Αυτό θα αποτελέσει καλή βάση για το νομοθετικό μας πλαίσιο. Ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία. Εύχομαι στην εισηγήτρια. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις αυτές. Θα παρακαλούσα τον πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, να πάρει το λόγο, τον ε, Διευθυντή για ε, την ψηφιακή κοινωνία, την κυρία Δέσποινα Σπανού να πάρει το λόγο και θα ήθελα να σας καλωσορί... να καλωσορίσω και τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Κατάινεν, Γιούρκη Κατάινεν. Uh, before end of our discussion, which is very, very interesting, cyber European σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν και δίνω το λόγο στην εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για να ακούσουμε ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα αυτό. Και κατόπιν θα δώσουμε το λόγο στην ε, εισηγήτρια. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την κοψή αυτή εισαγωγή και την ε, πίεση που ασκείται πάνω μου. Ε, κύριε Αντιπρόεδρε, σας ε, καλημερίζω. Έχουμε ε, εργαστεί υπό την ηγεσία του Επιτρόπου του Αντιπρόεδρου Κατάινεν στο θέμα αυτό, γι' αυτό γνωρίζει πολύ καλά το θέμα. Σας ευχαριστώ για την ε, πρότασή σας πάνω στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκθεσή σας προσέτει αξία στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όσον αφορά το πρώτο τμήμα, τα καθήκοντα της ΕΝΗΣΑ, βλέπουμε ότι η έκθεση αυτή συνεχίζει να ενισχύει ε, την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και γενικά βλέπουμε ότι κινείται εντός του ιδίου πνεύματος. Γι' αυτό ε, καλωσορίζουμε τη δουλειά που έχει γίνει. Όσον αφορά την πιστοποίηση, είναι κάπως πιο δύσκολα τα θέματα, διότι Βλέπουμε ότι γίνεται εδώ μια ειλικρινή προσπάθεια να επεκταθεί ε, περαιτέρω η δική μας πρόταση για ένα προαιρετικό σύστημα. Θα ήθελα να απαντήσω σε δύο παρατηρήσεις που έγιναν από ευρωβουλευτές κατά τη διάρκεια της συζήτησης αυτής. Καταρχάς, ο ρόλος των κρατών μελών. Στην πρότασή μας, τα κράτη-μέλη φυσικά παίζουν πρωτεύοντα ρόλο, συμμετέχουν σε αυτήν την νέα ομάδα που στόχο έχει τον πλήρη συντονισμό με την ε, ΝΙΖΑ για κάθε πρόγραμμα που προτείνεται και αξιολογείται. Το πρόβλημα είναι το να έχουμε ε, ένα επίπεδο έγκρισης πριν την αξιολόγηση ενός προγράμματος ε, μπορεί να έχει επιπτώσεις όσον αφορά τον χρόνο και τους πόρους που έχουν στη διάθεσή τους τα κράτη-μέλη κάθε πρόγραμμα ούτω ή άλλω εγκρίνεται με εκτελεστική πράξη, δηλαδή ούτω ή άλλω ψηφίζουν τα κράτη-μέλη κατά την ε, έγκριση. Υπάρχει λοιπόν ένα τέτοιο επίπεδο έγκριση ε, και καθ' όλη τη διάρκεια της ε, διαδικασίας. Το πρόβλημα με την πλήρη αξιολόγηση είναι ότι μπορεί έτσι να έχουμε καθυστέρηση στην ε, ένταξη στην αγορά των προγραμμάτων αυτών. Όσον αφορά τον ρόλο των ενδιαφερομένων, η μόνιμη ομάδα ενδιαφερομένων, η μόνιμη ομάδα stakeholders, είναι μια ομάδα που προτείνει ο Διευθυντής σύμφωνα με τους ε, κανόνες που ισχύουν αυτή τη στιγμή και που έχουν καθοριστεί στην ε, πράξη για την κυβερνοασφάλεια. Πιστεύω λοιπόν ότι θα είναι δύσκολο να μπορούμε να συγκεντρώσουμε εδώ εμπειρογνωμοσύνη για όλα τα θέματα και η έκθεση ε, πολύ σωστά αναφέρει τη δυνατότητα ομάδων εμπειρογνωμόνων ad hoc. Ο αναπληρωτής διευθυντής λοιπόν μπορεί να προτείνει δημιουργία ειδικών ομάδων για συγκεκριμένα προγράμματα κάτι που πιστεύουμε ότι επηρεάζει την αποτελεσματικότητα της πρότασής μας ε, είναι το θέμα της ε, έγκρισης. Ε, το να έχουμε την έγκριση των stakeholders πριν ψηφιστεί μια, ένα πρόγραμμα από τα κράτη-μέλη νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε. Δηλαδή πώς μπορούν να συμμετάσχουν οι ενδιαφερόμενοι χωρίς να καθυστερούν τη διαδικασία. Ε, ξέρω ότι εξήγησα το χρόνο μου ή έχω λίγο παραπάνω. Μου δίνετε λίγο ακόμα. Όχι. Νομίζω ότι αυτά είναι τα πιο βασικά θέματα και μία λέξη ακόμα. Εάν θέλουμε να αναθέσουμε περισσότερα καθήκοντα στην ΕΝΙΖΑ ε, όσον αφορά την πιστοποίηση, δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε ε, να τη δώσουμε και τους απαραίτητους πόρους. Ε, αυτή τη στιγμή έχουμε έγκριση μόνο για 14 επιπλέον άτομα. Ενώ η πιστοποίηση χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια από τον οργανισμό που είναι ήδη αρκετά μικρός. Εμείς την οδηγία την εγκρίναμε ε, αναθέτοντας πολλά καθήκοντα χωρίς όμως ε, την απαραίτητη πικοδότηση. Θα πρέπει να φροντίσουμε λοιπόν αυτά να πηγαίνουν μαζί, μαζί, να πηγαίνουν μαζί χέρι χέρι. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σπανού. Πολύ σημαντικές οι παρατηρήσεις σας και για την εισηγήτρια και για τους κοιόδη εισηγητές. Κυρία εισηγήτρια, σας παρακαλώ να συνοψίσετε τη συζήτησή μας. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες τις παρατηρήσεις σας και προτάσεις. Νομίζω ότι θα πρέπει να ε, ε, εργαστούμε πολύ αναλυτικά και να συνεχίσουμε την ε, συζήτηση με τους σκιώδεις εισηγητές και με οποιονδήποτε άλλο ενδιαφέρεται. Δεν χρειάζεται να αναφερθώ πάλι αναλυτικά στην πιστοποίηση. Ακούστηκαν πολλοί ενδιαφέρουσες ιδέες, ε, θα τις συνοψίσω όλες ε, και περιμένω τις τροπολογίες σας ε, με τη βάση των οποίων θα μπορέσουμε να δούμε πού μπορούμε να συμφωνήσουμε και πού όχι. Άλλωστε ο διάβολος στη λεπτομέρεια υπάρχει και θα πρέπει να λάβουμε κάποιες αποφάσεις. Θέλουμε αυτορύθμιση ή θέλουμε μια υποχρεωτική ρύθμιση. Όλα όμως τα θέματα αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Έχει να κάνει αυτό και με τα επίπεδα ασφαλείας και με τον ρόλο των κρατών μελών. Πολλά ερωτήματα αναπάντητα, τα οποία όμως πολύ ευχαρίστω θα εξετάσω στη συνέχεια με τους συναδέλφους. Είμαι βέβαιη ότι θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα καλό σύστημα, το οποίο θα πρέπει να είναι λειτουργικό, αποτελεσματικό και αυτό που υπογράμμισαν πολλοί συνάδελφοι εδώ πέρα θα πρέπει ε, να ε, συνάδει και με το ευρωπαϊκό πνεύμα που θέλουμε να βρισκόμαστε σε 10-15 χρόνια από τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια. Νομίζω ότι δεν υπήρχαν καν τόσες διαφωνίες όσες ε, περιμένατε πριν. Είναι καλύτερα λοιπόν τα πράγματα καλό σημάδι για σας, όμως ε, είναι ανοιχτή η συζήτηση, είναι όλοι ανοιχτή Η Σκιώδης, 26 Απριλίου είναι η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών, την Πέμπτη. Στις 12 το μεσημέρι. Πολύ σημαντικό θέμα. Και η ψηφοφορία στην Ήτρε στις 19 Ιουνίου. πολύ στενό χρονοδιάγραμμα. Καλή επιτυχία λοιπόν για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Και τώρα μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 5 της ημερησίας διάταξης. Καλωσορίζω τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Κατάινεν, εκ νέου. Είμαι Επίτροπος και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδιος για την απασχόληση, ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα. Πάρα πολύ σημαντικά θέματα αυτά για τους πολίτες και την οικονομία. Έχουμε μια αντιλαγή στο πλαίσιο του διαρθρωμένου διαλόγου. Και αν μου επιτρέπετε να πω ότι οι τρία θέματα είναι τα πιο σημαντικά για μας. Καταρχήν το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Βιομηχανικής Ανάπτυξης στην Άμυνα που είναι όλο καινούριο. Θέλουμε να ακούσουμε την άποψή σας ως Αντιπρόεδρο. έχοντας ε, φυσικά ε, και κατά νου και ε, τις απόψεις των 6-8 άλλων επιτρόπων. Επίσης υπάρχει ένα εκρεμές θέμα που αφορά την βιομηχανική πολιτική και άλλο ένα θέμα αφορά τα προγράμματα μετά το 2020 στο δικό σας ε, χαρτοφυλάκιο και υπό, το, υπό τις δικές μας Γιατί θέλουμε να ολοκληρώσουμε τον προπολογισμό για τα επόμενα 7 έτη. Θα ήθελα λοιπόν να σας ζητήσω να απαντήσετε σε αυτά τα ζητήματα, αλλά φυσικά και Μπορείτε να αναφέρετε και οποιοδήποτε άλλο θέμα εμπίπτει στις δικές σας αρμοδιότητες αλλά και στις δικές μας. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε και έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Πάντοτε είναι μεγάλη ικανοποίηση να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας για την ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση και τις επενδύσεις. Και φυσικά και πάνω στα θέματα που ανέφερε ο Πρόεδρος. Θα αναφερθώ στην αρχή στο θέμα των οικονομικών μεγάλων τάσεων που έχουν αντίκτυπο στην οικονομία μας αλλά και στις βιομηχανίες μας. Γιατί θα πρέπει να προσδιορίσουμε ποιες είναι οι κύριες τάσεις που θα αλλάξουν τον τρόπο που δημιουργείται η απασχόληση, η θέση εργασίας και που προκαλούν την ανάπτυξη αλλά και θέτουν προκλήσεις στη σημερινή κατάσταση γιατί δεν μπορούμε να βελτιώσουμε τη βιομηχανική μας ανταγωνιστικότητα ή να περιμένουμε μεγαλύτερη ανάπτυξη από τις επιχειρήσεις αν ε, δεν βρίσκονται στο μέσο αυτών των ε, κυρίαρχων τάσεων. Η ευρωπαϊκή οικονομία και η βιομηχανία αντιμετωπίζουν ε, τρεις παράλληλες προκλήσεις. Καταρχήν, ε, ταχύς τεχνολογικές ε, αλλαγές, παγκόσμια ανταγωνιστικότητα και την πρόκληση της βιωσιμότητας. Και Φυσικά δεν έχουμε μόνο αυτές τις προκλήσεις για την δική βιομηχανία, αλλά και για τη βιομηχανία παγκοσμίω. Θα πρέπει να παραδεκτώ επίση ότι οι πολιτικές που μπορεί να λειτουργήσαν πριν 20 χρόνια θα πρέπει να προσαρμοστούν για να λάβουμε υπόψη τις τάσεις ε, της ε, παγκόσμιας οικονομίας αλλά και των κοινωνιών μας. Κάτι για την ε, ψηφιοποίηση και για την ενεργειακή αποδυτικότητα, το χάρη, αλλά υπάρχουν και άλλα. Πιστεύω ότι μία από τις κυρίαρχες τάσεις στην παγκόσμια οικονομία θα είναι η κυκλική οικονομία, που ήδη καθίσταται η νέα πραγματικότητα. Δηλαδή η μετακίνηση από γραμμικά σε κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα συμβαίνει ήδη και ε, ε όσο μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι ε, σε πρώτη γραμμή, τόσο το καλύτερο για μας μακροπρόθεσμα. Επίσης ε, έχουμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα γίνει ε, κύριε Σπεκτής όταν θα έχουμε ε, την νομοθεσία που θα λαμβάνει υπόψη την κυκλική λογική και θα βοηθά τις επιχειρήσεις. Μία άλλη μεγάλη τάση και κινητήριο δύναμη είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Ενώ η Ευρώπη μπορεί να ήταν λιγότερο ενεργή από άλλου μέχρι τώρα στον τομέα αυτό, τώρα είμαστε αποφασισμένοι να επιταχύνουμε. Έχουμε ε, ταλέντο, έχουμε μια ισχυρή ερευνητική κοινότητα και ε, ισχυρά πρότυπα που θα προωθήσουν την διαλειτουργικότητα και θα παρουσιάσουν νέες λύσεις. Μπορεί να ρωτήσετε λοιπόν τι κάνει η Κομισιόν για όλα αυτά. Πώς μπορούμε να συνεργαστούμε για να διασφαλίσουμε ότι θα είμαστε στην ηγετική θέση σε ό,τι αφορά ε, τις κυρίαρχες τάσεις. Κατά τη διάρκεια της εντολής αυτής της Κομισιόν, η Κομισιόν ήδη υλοποίησε μια συντονισμένη και στρατηγική προσέγγιση και έχει φέρει αποτελέσματα στις προτεραιότητές της επενδυτικό σχέδιο, ε, στρατηγικές για την ψηφιακή γενιά αγορά, ενεργειακή ένωση, ένωση κεφαλαίου και θεματολόγιο για το εμπόριο. Βάσει των προτεραιοτήτων αυτών επικεντρωθήκαμε σε μεγάλα θέματα. Μία ένας από τους ε, τομείς αυτούς ε, ήταν και η ανταγωνιστικότητα της ε, βιομηχανίας. Μας ανοθήσαμε τη νέα στρατηγική για τη βιομηχανική πολιτική πέρσι. Ο ρόλος είναι να ενδυναμώσει τις βιομηχανίες, να προσαρμοστούν και να καινοτομήσουν, κυρίως σε τομείς όπως η ρομποτική, το δίκτυο των πραγμάτων, η τεχνητή νοημοσύνη, η βιοοικονομία, η άμυνα και νέα ενεργειακά συστήματα που ουσιαστικά ε, είναι φαινόμενα μιας νέας βιομηχανικής ε, εποχής. Ο ρόλος μιας επιτυχούς βιομηχανικής πολιτικής είναι να δημιουργήσει τις καλύτερες συνθήκες και να ενδυναμώσει τις ικανότητες ε, των επιχειρήσεων να προσαρμοστούν. Η Κομισιόν ως μέρος των προσπαθειών αυτή την εβδομάδα θα μια ανακοίνωση για να διασφαλίσει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα υιοθετηθεί στο επίπεδο εδώ ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλη την ευρωπαϊκή οικονομία. Η Κομισιόν θα συνεισφέρει αυξάνοντας τη χρηματοδότηση για την έρευνα στον τομέα, υποστηρίζοντας τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για την πρόσληψη των νέων τεχνολογιών και διασφαλίζοντας ότι θα υπάρχει και το κατάλληλο νομικό πλαίσιο. Σύμφωνα με την ε, στρατηγική της βιομηχανικής πολιτικής, και σύμφωνα με την ανακοίνωση για την τεχνητή νοημοσύνη, η Κομισιόν ε, επικαιροποιεί ε, και τη στρατηγική τη ε, που αφορά μέρο τη στρατηγική, της κυκλικής οικονομίας. Η προηγούμενη στρατηγική οθετήθηκε το 2012. Όπω αναφέραμε στην ανακοίνωσή μα για τη βιομηχανική πολιτική, θέλουμε τώρα να ξαναδούμε αυτή τη στρατηγική σε σχέση με του στόχου τη βιώσιμη ανάπτυξη. Γι' αυτό η Κομισιόν έχει αναθεωρήσει τα αποτελέσματα αποτελέσματα της προηγούμενης στρατηγικής και έχει ε, ε, ε ουσιαστικά εκφραστεί σχετικά ο κύριος Μοέδας τον περασμένο Νοέμβριο. Ε, κάναμε μια δημόσια διαβούλευση συνεχίζεται το έργο για να έχουμε ένα ευρύτερο όραμα για τη βιοοικονομία. Οποιοδήποτε feedback από το Κοινοβούλιο και ιδίω από την Επιτροπή ΙΤΡΕ θα είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτο. Η σημασία της βιοοικονομίας αυξάνεται ήδη σήμερα οι ε, βιομηχανίες ε, αυτές ε, παράγουν 3 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Είναι σημαντικές για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών. Έχουμε μακροπρόθεσμες ε, ε, συνδέσεις με την ε, χημική βιομηχανία και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε νέες ανταγωνιστικές λύσεις στην αγορά ενώ θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε του στόχου ε, τη δράση για την κυκλική οικονομία. Αυτή θα είναι μια καταστάση από την οποία θα κερδίσουν όλοι. Α πούμε, των προσπαθειών μα να προωθήσουμε την ανάπτυξη τη βιομηχανία στο μέλλον, θέλω να δράξω την ευκαιρία να αναφέρω ε, και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Βιομηχανική ανάπτυξη στην Άμυνα και τις ε, προετοιμασίε για τα προγράμματα μετά το 2020. Αυτό θα παρουσιαστεί από την Κομισιόν τις επόμενε εβδομάδε ό,τι αφορά την άμυνα. Είναι σαφές ότι η Ευρώπη θα πρέπει να απαντήσει στις διάφορες απειλές ασφάλειας που παρουσιάζονται αυτή τη στιγμή. Αναφέρονται σε υβριδικές απειλές ε, στην ε, τρομοκρατία ε, το να αυξήσουμε την συνεργασία είναι ο μόνο τρόπος να αντιμετωπίσουμε αυτές τις απειλές αποτελεσματικά και πιστικά. Γι' αυτό, αν αναπτύξουμε τη συνεργασία στην άμυνα, ε, αυτό θα παραμείνει στο επίκεντρο του μελλοντικού μας προβληματισμού. Ε, είναι σαφές ότι χρειάζεται περισσότερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Η αυτής, ε, συγγνώμη, έλλειψη αυτής της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών μπορεί να κοστίσει από 25 δισεκατομμύρια έως 100 δισεκατομμύρια ευρώ στους πολίτες. 30% των δαπανών θα μπορούσαμε ε, να το εξοικονομήσουμε μέσω της συνένωσης ε, των ε, διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων. Η Κομισιόν έχει δημιουργήσει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας με δύο σκέλη, ένα για την έρευνα και ένα για τις ικανότητες, προκειμένου να επιτρέψουμε κοινέ αποκτήσεις ε, πέρσι ε, έχουμε μία δράση για την έρευνα στην άμυνα και ήδη αυτό μας δείχνει ότι η συνεργασία είναι δυνατή, αλλά ε, είχαμε και μία πρώτη επιχορήγηση για ένα consortium που δημιουργήθηκε από 15 κράτη-μέλη. Σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη ικανοτήτων, παρουσιάσαμε έναν κανονισμό που θεσπίζει για το 2019 και το 2020 το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στην άμυνα για να ε, έχουμε την ανάπτυξη ικανοτήτων στην άμυνα. Ο κανονισμός αυτός τώρα είναι υποσυζήτηση μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Πιστεύω ότι στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ε, τριμερών διαλόγων θα βρούμε μία καλή λύση και για να προσδιορίσουμε τον όρο των επιλέξιμων οντοτήτων ε, και ε, πώς μπορούμε να έχουμε και συγκεκριμένες διατάξεις για να υποστηρίξουμε τις μικρές και μεσές επιχειρήσεις. Ε, υπάρχει ένα καλθόδες θέμα που αφορά τη χρηματοδότηση του προγράμματος. Είναι εντελώς αντίθετες οι θέσεις. Έχουμε 100% είναι η θέση του Κοινοβουλίου από ε, χρηματοδότηση από τα περιθώρια, πλήρης αναδιάταξη για το Συμβούλιο. Όμως ε, θα πρέπει το Κοινοβούλιο να δεχτεί να βρούμε ένα συμβιβασμό. Αξιότιμα μέλη κύριε Πρόεδρε, να πω δύο λόγια και για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2020 ήδη προετοιμαζόμαστε για τις ε, μελλοντικές συζητήσεις για το επόμενο πολιτές πλαίσιο. Στην ε, Κομισιόν εξεκολουθούμε να εκπονούμε κάποιες αποφάσεις. Είναι σημαντικό το μελλοντικό πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο να αντικατοπτρίζει τις πολιτικές μας φιλοδοξίες. Στο στάδιο αυτό δεν μπορώ να αναφέρω λεπτομερίες για τις μελλοντικέ προτάσεις, όμως υπάρχουν ε, κάποια πράγματα που είναι σαφή και καθολικά. Καταρχήν είναι σαφές ότι η Ευρώπη θα πρέπει να συνεχίσει να επενδύει σε τομείς όπου είναι υψηλή προσθέμενη εξή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε έρευνα, ε, καινοτομία και ηγετική θέση στην τεχνολογία. Αυτές πρέπει να είναι προτεραιότητες για τον προπολογισμό. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε βέβαια ε, και τους περιορισμούς του προπολογισμού που προκύπτουν και από το Brexit. Θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα με λιγότερα και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε όσο δυνατόν μεγαλύτερη μόχλευση στον προπολογισμό της Ένωσης. Γι' αυτό ε, αναπτύσσουμε την έννοια του ε, Ταμείου για τις επενδύσεις Invest in You Fund. Θέλουμε να προωθήσουμε αυτή την προσέγγιση περαιτέρω στο νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Όμως η μεγαλύτερη διαφορά αυτή τη φορά είναι ότι δεν θα πρόκειται για κάτι ad hoc, δηλαδή θα έχουμε τον προπολογισμό και θα το κατανοούμε σε άλλους σκοπούς, αλλά θα έχουμε μια πιο διαρθρωμένη προσέγγιση η εφαρμογή των φιλόδοξων πολιτικών της Ένωσης, ε, πλαστικά, ενέργεια, κλίμα, απαιτούν σημαντικές επενδύσεις. Αυτές οι επενδύσεις ε, δεν μπορούν να, δοθούν, να γίνουν μόνο από το δημόσιο τομέα. Γι' αυτό αναπτύσσουμε την ε, έννοια ε, κάποιων ε, χρηματοδοτικών εργαλείων όπως είναι το ΕΦΣΙ, το οποίο θα αποτελέσει ένα μηχανισμό χρηματοδότησης πολλαπλών πολιτικών. τους χάρη θα έχουμε ε, χρηματοδότηση περισσότερο με λιγότερα αυξάνοντα τη μόχλευση. Μόνο αυτή η ε, προσέγγιση μπορεί να αυξήσει τι δυνατότητε χρηματοδότηση. Αν ε, επιλέξουμε ή προσέξουμε να σε δημόσια κονδύλια, δεν θα πετύχουμε του στόχου. Επίση, θα πρέπει να έχουμε ενίου κανόνε για τα προγράμματα. Η σημερική κατάσταση δεν είναι βέλτιστη. Έχουμε αρκετού χρηματοδοτικού μηχανισμού που αναφέρονται στον ίδιο στόχο παραδείγματο χάρη 7 διαφορετικού μηχανισμού που αφορούν τι μικρέ και μεσαίε επιχειρήσει. Ένα μηχανισμό ε, θα μπορούσε να είναι πιο ελκυστικό πολιτικά, θα αύξανε την διαφάνεια και την προβολή τη Ευρωπαϊκή ε, Ένωση καθώς ε, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και σε αυτό το οίκο πρέπει να πω τι δεν σκοπεύουμε να κάνουμε. Να είμαι σαφής. Ουσιαστικά εδώ δεν πρόκειται για φαρπαγή εξουσίας το αντίθετο ε, στην ε, Κομισιόν ε, ή σε κάποιες επιτροπές δεν θα αφαιρεθούν οι αρμοδιότητές τους. Το αντίθετο θα συνεχίσει να υπάρχει χρηματοδότηση. Μόνο η διαχείριση των δημοσιονομικών διατάξεων θα συνενωθούν. δεν ε, έχουμε εδώ αντίθεση με κάποιους μηχανισμούς που βασίζονται σε τάσει. Θα πρέπει να έχουμε συμπληρωματικά εργαλεία θα χρησιμοποιηθούν μόνο ε, σε τομεί όπου υπάρχει κενό στην αγορά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ε, και ιδιωτικά κεφάλαια αυξημένος αντίκτυπος στο να πετύχουμε μεγαλύτερη μόχλευση θα μας οδηγήσει στο να ε, χρησιμοποιήσουμε ε, το Ευρωπαϊκό ε, Ταμείο, το ΕΣΥΦ, με άλλα προγράμματα. Για να μπορεί να υπάρξει αυτός ο μηχανισμός χρειάζονται ενιαίοι κανόνες δεν ε, θα κάνουμε πιο πολύπλοκη τη σημερινή κατάσταση. Θέλουμε να απλωστεύσουμε. Τα σημεία αναφοράς ε, θα είναι ε, ουσιαστικά τα προγράμματα με τους ε, λιγότερο πολύπλοκους κανόνες, όχι το αντίστροφο. Αξιότιμα μέλη. Ήθελα να πω κάτι, μάλλον σκόπευα να πω κάτι για το εμπόριο, αλλά θέλω να αφήσω περισσότερο χρόνο για τη συζήτηση. Το προηγούμενο Σάββατο μπορέσαμε να υπογράψουμε μια συμφωνία με το Μεξικό, επομένως έχουμε τώρα μια σύγχρονη συμφωνία εμπορική και με το Μεξικό και με τον Καναδά και δεν πρόκειται για σύμπτωση. Υπάρχουν πολύ καλοί λόγοι να είμαστε ικανοποιημένοι γιατί είναι ένα σημαντικό εργαλείο αυτό για τη βιομηχανία και για να μπορέσουμε να πουλήσουμε καλύτερα τη γνώση μας και τα προϊόντα μας. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρόεδρε. Ναι, υπάρχει και το θέμα των εμπορικών δυνατοτήτων με, με τη Βόρεια Αμερική βέβαια. Δεν είναι τα πράγματα όπως ε, τα είχαμε κατά νου πριν από μερικά χρόνια, αλλά είναι ένα θέμα παρεμφερές. Λοιπόν, τώρα, εκ μέρους των πολιτικών ομάδων θα παρέμβουν κάποιοι ομιλητές. Από το ΕΛΚ πρώτα, ο κύριος Έλερ έχει το λόγο. Έχω και κάποια πρακτικ... ένα πρακτικό ερώτημα από τον κύριο Κατάνη. Αναφερθήκατε στη βιομηχανική πολιτική και στη σημασία καινοτομία. Ε, εάν δούμε όμω τα διάφορα στοιχεία, διαπιστώνουμε ότι ο τομέας ο οποίος αυξάνεται περισσότερο αυτή τη στιγμή είναι ε, ο βιομηχανικός ε, ο οποίος δεν καλύπτει τον συνάδελφο την κυρία Μπιανκόφσκα 12,9% είναι η αύξηση και αυτό ισχύει εδώ και 10 χρόνια. Τι θα κάνετε λοιπόν με την πρόταση αυτή του Κοινοβουλίου για τη συγκεκριμένη βιομηχανία, τις δημιουργικές, το νομέα της δημιουργίας, τη δημιουργική βιομηχανία. Στο Συμβούλιο έχει αποφασιστεί 3% του ΑΕΠ ε, να πάει στην καινοτομία. Τα στοιχεία όμως τώρα είναι 1,9%, 2%, ε, κάτω από το 2%. Το θεωρητικό στοιχείο που προκύπτει από τη συμμετοχή του κλάδου, του, του, ευρωπαϊκού προπολογισμού και των κρατών μελών είναι 195 δισεκατομμύρια ευρώ το 3%. Το ερώτημα είναι, εφόσον το Κοινοβούλιο είχε προτείνει 120 ε, δις που δεν φτάνει καν στον στόχο τον, τη φιλοδοξία την αρχική. Τώρα μας λένε ότι ε, πάμε ακόμα πιο κάτω. Ότι κατεβαίνει ο πύχης. Ποιες είναι λοιπόν οι προσδοκίες από αυτού. Και τελευταίο ερώτημα. Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά μέσα, στο πρόγραμμα πλαίσιο ε, ήταν ε, τα πιο ευέλικτα εργαλεία αυτά τα οικονομικά. Αφορά το R&D, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις πιο μικρές επασπτωσιοντότητες ε, και οι κανόνες είναι και πλέον ευέλικτοι γι' αυτό το, το μέσο. Ε, ενδεχομένως επειδή το Κοινοβούλιο δεν είχε αρκετό λόγο ή επειδή η Κομισιόν δεν είχε τόσο λόγο, ε, είναι πάντως ένα πολύ ευέλικτο εργαλείο. Και τώρα το εγγράφουμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ένα, ε, ένα σετ κανόνων για όλους ή αφήνουμε την ευελιξία των ε, μικρότερων μέσων, μικροματοδοτικών μέσων στην ισχύα, όπως, η ε, όπως το μέσο Ίνοφιν, Είναι σημαντικό να το γνωρίζουμε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες, η κυρία Καμπεθόν Ρουίθ. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Ε, κύριε Πρόεδρε, συγχαρητήρια για τη συμφωνία με το Μεξικό που όντως ήταν απαραίτητη και σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω ένα συγκεκριμένο ερώτημα να σας θέσω. Έχει να κάνει με το τη δυνατότητα ε, της ε, ε, παρασκευής φαρμάκων γενώσιμων όσο ισχύει το FPC. Ε, σύμφωνα με τους κανόνες που έχουμε, τα στοιχεία που έχουμε μάλλον, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαπιστώνουμε ότι έχει υπάρξει μετακατάσταση των επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς ε, εδάφη, προς, προς χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί εδώ δεν μπορούν να παρασκευαστούν. Ταυτόχρονα υπάρχει ένα θετικό αντίκτυπος, θα υπήρχε θετικό αντίκτυπος, εάν δεν υπήρχε πλέον αυτή η προστασία. Ε, όσο ισχύει η πατέντα, το δίπλωμα ευρωστεχνία. Δεν, δεν, δεν είναι θέμα πνευματική διοκτησίας, είναι ένα θέμα πολιτικό. Ε, θέμα βιομηχανικής πολιτικής. Θα ήταν λοιπόν θετικό αυτό, όχι μόνο για να μπορέσουμε να εξάγουμε, ε, αυτό είναι βέβαιο ότι θα ήταν ε, θετικό, ε, θα πρέπει η Κομισιόν να πάρει τα απαραίτητα μέτρα για να γίνει αυτό πραγματικότητα. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να μελετήσει τη δυνατότητα αυτή η Παρασκευή να επιτρέπεται έτσι ώστε να μπορεί να τεθεί στην εμπορία, σε εμπορία στην αγορά των γενοσύμων μόλις τελειώσει η περίοδος προστασίας του διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Γιατί όπως λέει μια μελέτη το 2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα αύξανε θα αυτό σημαντικά την εξοικονόμηση των ε, συστημάτων υγείας. Ε, μιλάμε για 15 δις το χρόνο. Αυτή η καθυστέρηση των 6 μηνών από τη στιγμή λοιπόν που θα λήξει το Τμήμα ευρωτεχνία, όσο του έχουμε τα επαρκή γενώσιμα για να μπορέσουμε να τα ε, εισάγουμε στην αγορά, ε, αυτό σημαίνει ε, μια απώλεια σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα εξοικονόμησης. Ε, σας, σας, σας, έλεγα λοιπόν ε, να, παρθ, να τα απαραίτητα αναμορφωτικά μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή έτσι ώστε η ευρωπαϊκή βιομηχανία να μην με, οδηγείται στη μετεγκατάσταση και να μπορεί ε, να παράγει γενώσιμα εδώ. Διότι υπάρχουν άλλες χώρες όπως η Ινδία και η Κίνα που αυτή τη στιγμή μας έχουν προσπεράσει. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Από το ECR τώρα ο κύριος Τοσανόφσκι έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ένα ερώτημα μόνο. Είπατε στην εισαγωγή σας, αναφερθήκατε στις τρεις βασικές τάσεις και εγώ συμφωνώ, ε, αναφερθήκατε και στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Αναρωτιέμαι όμως, αυτή η προσπάθεια να εξευρεθεί μια διοικητική λύση μήπως τελικά ε, πλήττει την ανταγωνιστικότητα, μήπως ε, δίνουμε ιδιαίτερο, ιδιαίτερη έμφαση στον διοικητικό έλεγχο και στον στατιστικό έλεγχο. Εδώ να αναφέρομαι στην Ενεργειακή Ένωση. Ε, ήταν μια ενδιαφέρουσα ιδέα αρχικά. Ήταν έτσι μια εμπνευσμένη πρωτοβουλία. Όμως αυτή τη στιγμή φτάνουμε σε ένα σημείο όπου περιορίζουμε την τεχνολογική ουδετερότητα, ε, γίνονται αξιολογήσεις στατιστικές ε, που πάνε στο, το 2050, δηλαδή μιλάμε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, αντί να κινηθούμε προς τα εκεί, ε, προς το δρόμο που αναφέρατε εσείς, ε, καινοτομία, έρευνα, στήριξη της έρευνας και της εκπαίδευσης, χωρίς ε, να αποκλείουμε εκ των προτέρων κάποιες τεχνολογικές λύσεις ε, που θα μπορούσαν ενδεχομένως να δημιουργήσουν μεγαλύτερη αγωνιστικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ο κύριος Τάλιτσκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλό απόγευμα κύριε Αντιπρόεδρε. Χαίρομαι που βρίσκεστε εδώ. Δεν έχω ερωτήσεις για ένα βασικό λόγο ε, πρέπει να αποχωρήσω να πάω σε μια άλλη συνεδρία και θα ήταν αγενές να μην περιμένω την απάντησή σας. Κάποιες παρατηρήσεις όμως. Νομίζω ότι πολύ σωστά μιλήσατε για την ε, ψηφιακή οικονομία. Θυμάμαι τη μέρα που είχατε παρουσιάσει τη δέσμη μέτρων ε, στην Ολομέλεια και ήταν πολύ σωστή η προσέγγιση της ε, Κομισιόν. Ήμουνα σκιώδης ε, στην ε, Ήτρε σε δύο από τα θέματα αυτά, αλλά η μεγάλη πρόκληση είναι να εξετάσουμε πώς μπορούμε να πετύχουμε την αλλαγή στα κράτη-μέλη, διότι αλλάζουμε νοοτροπία πολύ αργά σε κάποια κράτη-μέλη. Ίσως στο μέλλον το Ευρωπαϊκό Τομείο Στρατηγικών Επενδύσεων να μπορέσει να παίξει σημαντικό ρόλο, όχι μόνο όσον αφορά ε, το ποσοστό που θα δοθεί στην κυκλική οικονομία, αλλά η Είπατε ότι θέλετε να σκεφτείτε τις προτεραιότητες. Ίσως να έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε το θέμα αυτό στο μέλλον. Όσον αφορά το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, στο οποίο αναφερθήκατε, και όπου είπατε ότι θέλετε να συζητήσετε τις προτεραιότητες, ε, ένα βασικό θέμα εδώ είναι οι προϋποθέσεις. Θα πρέπει να εισάγουμε προϋποθέσεις ώστε να προσπαθούμε να πετύχουμε ακριβώς τους στόχους που αναφέρατε. Το αν οι προϋποθέσεις αυτές θα είναι θετικές ή αρνητικές, το σημαντικό είναι να λειτουργήσουν καλά. Αρκετά κράτη-μέλη θα πρέπει να εισάγουν μεταρρυθμίσεις. Ε, δεν το αναφέρατε αυτό, νομίζω όμως ότι είναι ένα θέμα κλειδί και πιστεύω ότι οι προϋποθέσεις ε, θα μπορέσουν να παίξουν σημαντικό ρόλο εδώ και όσον αφορά τους πόρους που έχουν στη διάθεσή τους. Μια τελευταία παρατήρηση. Όσον αφορά το διοικητικό άχθος, έχουμε πετύχει πρόοδο, έχουμε δει αλλαγή νοοτροπίας ε, και εντό τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κάπως λιγότερο εδώ στο Κοινοβούλιο, αλλά συνεχίζω να είμαι αισιόδοξο. Δεν θα πρέπει όμως ε, να ε, απατώμεθα. Το διοικητικό άχθος συνεχίζει να αυξάνεται, ούτε το έχουμε μειώσει, ούτε καν το έχουμε σταθεροποιήσει. Θα πρέπει λοιπόν να εισάγουμε εργαλεία ώστε να σταθεροποιηθεί να μείνει στάσιμο. Παρά τι προσπάθειε Ευρωπαϊκή Επιτροπής συνεχίζει να αυξάνεται. Όσον αφορά τα θέματα άμυνα. Θα συμφωνήσω, δεν είναι εύκολο καθότι δεν έχουμε κοινή πολιτική άμυνα ε, και επειδή δεν γνωρίζουμε πόσο πολύπλοκο θα είναι το θέμα, αναφερθήκατε όμω στι δημόσιε συμβάσει και αυτό σίγουρα μπορεί να αποτελέσει προτεραιότητα. Η έρευνα αποτελεί δεύτερη προτεραιότητα δεν βλέπω να γίνονται πολλά στον βιομηχανικό τομέα. Ε, όσον αφορά τις ε, μεταφορές, γενικά το θέμα των υποδομών μπορεί να αποτελέσει ε, σημείο το οποίο θα πρέπει να εξετάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα κλείσω εδώ για λόγους περιορισμένου χρόνου. Πολύ ευχαριστώ όμως. Θα συνεχίσουμε να προβληματοζόμαστε μαζί πάνω στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ κύριε Λόπες από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστούμε κυρία κατάνια για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Αναφερθήκατε σε κυριαρχές τάσεις ε, και σε πολύ μεγάλες προκλήσεις. Δυστυχώς υπάρχει όμως αναθεμελιώδης ε, και δεν σχολιάσατε καθόλου το θέμα αυτό. Αφορά το θέμα της συμμετοχής των πολιτών σε όλο αυτό το μέλλον που μας ε, εκθέσατε. Όχι μόνο δεν εξελίψαμε τα παλιά χάσματα, αλλά ούτε δίνουμε μια ικανοποιητική απάντηση στα νέα χάσματα που λαμβάνουν χώρα αυτή τη στιγμή, υπάρχουν το σχάλι, στην ψηφιακή εποχή, στα νέα βιομηχανικά μοντέλα. Είναι πολύ απλή η ερώτησή μου. Πώ θα είναι η κοινωνία που θέλουμε να ζήσουμε. Η παγκόσμια ανταγωνιστικότητα δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία για την ε, επιδείνωση των δικαιωμάτων και αυτό ακριβώ συμβαίνει στην Ευρώπη εδώ και χρόνια πώς ε, θέλουμε να οικοδομηθεί αυτή η Ευρώπη και δεν μπορεί να γίνει εκβιομηχάνηση του κέντρου εις βάρος της αποβιομηχάνησης της περιφέρειας και αυτό ακριβώ σημαίνει με το Ταμείο Εύσης Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων καλύπτονται οι ανάγκες του κέντρου και υπάρχει αποβιομηχάνηση στην περιφέρεια και φυσικά ο μειωμένο προπολογισμό δεν συνάδει με τις αυξανόμενε φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Ένωση, Το να προσφύγουμε στην ιδιωτική χρηματοδότηση αποτελεί λαχιοφόρο αγορά, ε, ενώ εμεί ζητάμε την υλοποίηση ε, των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει και επιχειρήσει. Ποιο είναι ο βαθμό ε, της υπευθυνότητα και των επιχειρήσεων και του βαθμού υλοποίηση των δεσμεύσεων αυτά που μας παρουσιάσατε σήμερα πράγματι θα είναι η απάντηση στο 57% των νέων Ευρωπαίων που δηλώνουν ότι αισθάνονται αποκλεισμένοι από την εργασιακή και οικονομική και κοινωνική ζωή και αποτελούν το μέλλον αυτής της Ευρώπης. Ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις σας. και τώρα να περάσουμε στους υπόλοιπους ομιλητές. Η κυρία Γκροστέτ καταρχήν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Αντιπρόεδρο της Κομισιόν που ήρθε να μας μιλήσει για όλα αυτά τα σημαντικά θέματα ε, την εξέλιξη της κοινωνίας αυτή τη στιγμή ζούμε σημαντικές ανατροπές. Συμφωνώ απόλυτα με όσα είπατε σε ό,τι αφορά την κυκλική οικονομία, την τεχνητή νοημοσύνη. Πράγματι, θα πρέπει να ασχοληθούμε επιτέλους, γιατί σημειώνεται μεγάλη πρόοδος σε άλλες υπήρους και Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσδώσουμε το απαραίτητο πλαίσιο, αλλά και να καθησυχάσουμε κάπως τους συμπολίτε μας που μερικές φορές ανησυχούν ε, με αυτές τις εξελίξεις. Ε, εγώ θεωρώ ότι μπορεί να είναι πολύ ενθουσιώδης, αλλά μπορούμε να κατανοήσουμε ότι κάποιοι συμπολίτε μας ανησυχούν πάρα πολύ. Και ε, ίσως θα πρέπει να προβληματιστούμε σε κοινωνικό επίπεδο για το θέμα της εξέλιξης της τεχνητής νοημοσύνης. Φυσικά θα ήθελα να σας πω ότι σας υποστηρίζω πλήρως για την ε, πολιτική άμυνας και την πολιτική διαστήματος. Άκουσα ότι είπατε ότι ε, το Κοινοβούλιο πρέπει να κάνει μια προσπάθεια για τον προπολογισμό της άμυνας, αλλά εγώ ζητώ και το Συμβούλιο να κάνει την ίδια προσπάθεια. Δύο είμαστε εδώ σε μια διαπραγμάτευση. Το Κοινοβούλιο είναι πράγματι απολύτως αλληλέγγυο και ενωμένο για αυτό το Ταμείο Άμυνας. Ε, τον προϋπολογισμό πράγματι είναι εντελώς ε, αντιδιαμετραστικά αντίθετε οι θέσει, όμω ε, μη ζητάτε μόνο από το Κοινοβούλιο να κάνει προσπάθειε και το Συμβούλιο πρέπει να κάνει προσπάθειε. Επίση, ε, θα πρέπει να κάνει προσπάθειε για να κατανοήσει τι εγγύσει που θέλει το Κοινοβούλιο να ισχύουν για τα κριτήρια επιλεξιμότητα. σω θα το ξανασυζητήσουμε όμω. Στη συνέχεια. Έχετε λοιπόν πολλές φιλοδοξίες, ε, βεβαίως και εμείς τις συμμεριζόμαστε, όμως θέλω να σας θέσω το εξής ερώτημα. Υπάρχει ομάδα εργασία με επικεφαλή στον Πασκαλαμή και πρότεινε να διπλασιαστούν τα μέσα για το επόμενο ε, πρόγραμμα πλαίσιο. Ο αρμόδιο επίτροπο για τα ψηφιακά μα είπε ότι θα πρέπει να διπλασιάσουμε τον προπολογισμό. Για τα ψηφιακά τώρα μα είπατε πρέπει να τα καταφέρουμε καλύτερα με λιγότερα χρήματα. Θα πρέπει κάποια στιγμή να έχουμε το θαρρο να θέσουμε τα πράγματα επιτάπητο και να ρωτήσουμε το Συμβούλιο αν ε, θέλει ε, πραγματικά να ε, ακολουθήσει ε, τον εξυγχρονισμό ε, αυτό τον αιώνα ή αν θέλει να καθυστερούμε σε όλους τους τομείς και φυσικά θα έχουμε όλο ένα και μικρότερη επιρροή ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, λοιπόν, τι πιστεύετε για τα συμπεράσματα του Πασκάλ Λαμή και τι θα κάνετε σε σχέση με τον προβλησμό και τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Βαν Μπρέμπτ. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τον κύριο Επίτροπο που είναι εδώ και που μας έκανε την εισαγωγή του. Τρεις ερωτήσεις, θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομη. Καταρχάς, ε, φυσικά στηρίζω τη στήριξη που παρέχετε εσείς ε, στην κυκλική οικονομία. Νομίζω ότι όλοι εδώ στην Επιτροπή μας ε, θα συμφωνήσουν ότι αυτό αποτελεί ζωτικό τμήμα της μελλοντική μας οικονομίας. Την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο υιοθετήσαμε την τελική δέσμη μέτρων. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε το λάθος να θεωρήσουμε ότι αυτό είναι ολοκληρωμένο πακέτο. Ε, λείπουν ακόμα κάποια θέματα και ένα από αυτά είναι η προσέγγιση του οικολογικού σχεδιασμού, η οποία, ο οποίος ε, στο παρελθόν ήταν πολύ επιτυχής ε, ώστε να έχουμε αποδοτικά προϊόντα. Τώρα όμως ε, θα πρέπει να έχουμε ε, σφαιρική οπτική στον τομέα αυτών. Ε, νομίζω λοιπόν ότι η σχετική πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αποτελέσει πολύ καλό κλείσιμο της δέσμης μέτρων αυτής. Ε, δεύτερον, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Γνωρίζετε ότι για την δική μας πολιτική ομάδα ήταν και συνεχίζει να είναι πολύ σημαντικό το να διασφαλίσουμε το βασικό επίκεντρο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων να είναι η βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Όταν μιλάμε για την βιομηχανία του μέλλοντος, ε, ε, θα πρέπει να δώσουμε και μια όθηση στη βιομηχανία μας ε, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στο μέλλον. χωρίζουμε τις βιομηχανίες, λέμε ότι αυτές είναι ε, αηφόρες, ε, οι άλλες είναι κλασικές. Όχι, θα πρέπει να έχουμε μια σφαιρική εικόνα. Θα πρέπει να φροντίσουμε να συνδυάσουμε τη βιωσιμότητα με τις άλλες πτυχές ε, και θα ήθελα πολύ να ακούσω τους προβληματισμούς σας πάνω στο θέμα αυτό όσον αφορά δηλαδή τη ματιά μας προς το μέλλον. Και κάτι ακόμα, αναφερθήκατε στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο με αρκετά θολούς όρους. Ε, ναι, φυσικά κάποια πράγματα απομένουν ακόμη να γίνουν και ε, το βασικό επίκεντρο θα πρέπει να είναι η καινοτομία, αλλά και άλλα θέματα κοινοτικά, ε, κοινωνικά, συγγνώμη, ταμείο συνοχής κλπ. Ωραία τα συνθήματα, όμως όλοι αναζητούν ε, λύσεις από την Ευρώπη, ε, αλλά το να κάνουμε περισσότερα με λιγότερα είναι ωραίο σύνθημα, αλλά δύσκολο. Θα πρέπει λοιπόν ε, να στηρίξετε το Κοινοβούλιο στις εργασίες του και ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις και το Συμβούλιο να γνωρίζει επίσης τον σχετικό προβληματισμό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο επόμενος ομιλητής τώρα. Η κυρία Νίμπλερ. Äh, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίασή σας. Αναφερθήκατε στις ε, βασικές τάσεις ε, στην οικονομία και αναφερθήκατε και τις ε, στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να ανταποκριθεί στις τάσεις αυτές έχω την εξής ερώτηση. Εάν ε, είναι να ε, αξιολογήσετε τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πού βρισκόμαστε όσον αφορά αυτές τις βασικές τάσεις. Πού στεκόμαστε αυτή τη στιγμή. Και κατά συνέπεια, σε ένα χρόνο έχουμε ευρωεκλογές ε, και το τέλος της θητείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, τι θα έχουμε να παρουσιάσουμε στους πολίτες μας τότε. Αυθόρμητα, ποια θα ήταν η απάντησή σας, ε, ποια είναι τα τρία βασικά θέματα, ποια είναι τα βασικά μηνύματα που μπορούμε να μεταφέρουμε στους πολίτες μας ε, όσον αφορά τον οικονομικό τομέα. Θα με ενδιαφέρει πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο κύριος Μαρτά έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Εδώ, εδώ αριστερά. Που μας παρουσιάσατε ποια είναι η άποψή σας, ποια είναι το όραμά σας για την ευρωπαϊκή μηχανία ε, του μέλλοντος. Ε, όλοι από το Στρασβούργο επιστρέφουμε, δεν ξέρω αν ήσασταν και εσείς. Ο κύριος Γιούγκερ είπε κάτι ενδιαφέρον. Ε, έτσι μας εξέπληξε κάπως, αλλά ήταν ενδιαφέρον. Είπε ότι δεν θέλει μια Ευρώπη Ο κύριος Μακρόν μίλησε για μια κυριαρχία ευρωπαϊκή ε, που να προστατεύει τους Ευρωπαίους διότι ο κόσμος βράζει. Υπάρχει όμως και ένα άλλο σημείο που βράζει ο κόσμος. Θα ήθελα να αναφερθώ για τους εσωτερικού κανόνες ανταγωνισμού. Θα αναφερθώ σε ένα ταμπού, ίσως για σας, ε, ίσως να είναι ε, και το προπατορικό αμάρτημα, τι να πω. Είναι ο ορισμός του κατάλληλου γεωγραφικής αγοράς. Όταν μια επιχείρηση έχει 30% του μερίδιου, αγορά μια βιομηχανία, θεωρούμε ότι έχει τις θέση και η, η Κομισιόν την, την υποχρεώνει να καταλήψει ε, κάποιες εγκαταστάσεις, όπως η ArcelorMittal. Εδώ λοιπόν ε, προσφέρουμε ε, γενναιόδωρα στο διεθνή ανταγωνισμό ε, κάποιες, ε, κάποιον κλάδο όπως η Ρωσία, όπως η Κίνα που δεν σέβονται βεβαίως τις, ε, τα κριτήριά μας, τα περιβαλλοντικά, τα κοινωνικά, δεν έχουν κανόνες ανταγωνισμού στο εσωτερικό τους οι ίδιοι. Ταυτόχρονα η Κίνα ε, στον τομέα του αλουμινίου, στον τομέα των σειροδρόμων έχει 50% του παγκοσμίου μερίδιου αγοράς, πάνω από 60% στην Ασία. Το ερώτημα μου είναι απλό κύριε Επίτροπε πότε θα αντιληφθούμε ότι αυτή τη στιγμή ο ανταγωνισμός είναι παγκοσμιοποιημένος και πότε θα τολμήσετε να πείτε ότι πρέπει να αλλάξουν οι συνθήκες μας. ότι καλό είναι να έχουμε κάποιες ιδέες για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Θα πρέπει όμως να μην καταστρέφουμε τους υπάρχους, τις υπάρχουσες θέσεις απασχόλησης. Αυτό που με ενοχλεί εμένα είναι ότι προσπαθείτε εδώ να μας πείτε ότι πρέπει να δημιουργήσουμε νέα εργαλεία χωρίς όμως να ανανεώσουμε τα υπάρχοντα εργαλεία τα οποία δεν είναι πλέον κατάλληλα. Και εδώ Ξέρετε πολύ καλά ότι οι εισαγωγέ θα έρθουν από μια περιοχή εκτός Ευρώπη. Εμείς εδώ προσφέρουμε, θυσιάζουμε το, την βιομηχανία μας. Να φανείτε λοιπόν καινοτόμοι, γενε, γενναιόδοροι και να αλλάξετε τη συνθήκη έτσι ώστε να ξαναδούμε τους κανόνες του ιστορικού ανταγωνισμού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ναι, εδώ αναφέρεται φαντάζομαι σε κάποιου εθνικούς πρωταθλητέ ε, και πώ θα αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα στο μέλλον. Είχαμε ένα τέτοιο πρόβλημα με εθνικούς πρωταθλητέ ε, και στον τομέα της ενέργεια. Και υπήρχε ένα θέμα, ε, το θέμα της ιδιοκτησίας του ownership unbundling, το οποίο μπορούσε να βοηθήσει στην τέτοια περίπτωση. Η κυρία Βίρινγκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε κύριε Κατάινεν. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ. Ένα ερώτημα έχω μόνο για σας. Στην ΙΤΡΕ, στην Επιτροπή ΙΤΡΕ, ετοιμαζόμαστε για το επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο. Ως φιλελεύθερη, εγώ πιστεύω πραγματικά στις επενδύσεις, στην καινοτομία και την έρευνα. Αυτές εξασφαλίσουν την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα μακροπρόθεσμα στην Ευρώπη. Από εκεί και πέρα όμως θα ήθελα μια πραγματική αύξηση στο FP9 e αύξηση του προπολογισμού, όπως είπε και ο συνάδελφος. Πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βλέπει την κατανομή ε, του προπολογισμού για τον τομέα της έρευνας και μετά το 2020. Ευχαριστώ. Ο κ. Κόχλιτσεκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι εδώ λίγο αριστερά σας. Κύριε Επίτροπε, ναι, εδώ είμαι. Έχω κάποια ερωτήματα να σας θέσω. Η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να καταλάβουμε ότι σε μια σειρά τομείς και το είπαν και οι συνάδελφοι, αναφέρθηκαν τρεις χώρες, ε, ε στις Ηνωμένες Πολιτείες ε, έχουμε αθέμητο ανταγωνισμό, κλασικό αθέμητο ανταγωνισμό, ε, στον τομέα της κατανάλωσης ε, ο κλασικός του ανταγωνισμό, έχει να κάνει με το Μπαγκλαντέ, το Πακιστάν, ε, στην Νοτιοανατολική Ασία. Ε, πώς πιστεύετε ότι μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Εάν στην Τσεχία, που δεν είναι από τι πιο ακριβές χώρε τη Ένωση, εάν θέλει κάποιος ε, να κατασκευάσει ε, ένα μηχανάκι όπως αυτά που εισάγουμε από την Κίνα, μόνο τα εξαρτήματα είναι, κοστίζουν τριπλάσια. Α, τριπλάσια από το έτοιμο μηχανάκι που αγοράζει κανείς από την Κίνα. Πώς μπορούμε λοιπόν να προστατεύσουμε πώς μπορούμε να προστατεύσουμε αυτούς τους βιομηχανικούς κλάδους. Επίσης αυξάνεται το διοικητικό άχθος. Πώς ε, θα μπορέσουμε στον τομέα της, ε, της επιστήμης, της έρευνας, ε, των νέων τεχνολογιών, πώς μπορείτε να αποτρέψετε οι οδηγίες ε, να μας ξεπεράσουν τελείως. Φαντάζομαι ότι έχετε ένα σχέδιο απλούστευσης ό,τι αφορά τις διάφορες οδηγίες, έτσι ώστε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έτσι ώστε ο μικροεπιχειρηματίας να μπορέσει να βγάλει άκρη, εάν θέλουμε να τον βοηθήσουμε. Επίσης ε, η Κίνα κάνει πιο αυστηρούς ε, τους κανόνες ό,τι αφορά την εισαγωγή των πλαστικών ε, αποβλήτων και αυτό δημιούργησε μεγάλη αναταραχή και στην Ευρώπη. Έχουμε προγράμματα για να ενθαρρύνουμε την μεταποίηση όχι μόνο του πλαστικού τα μπουκάλια, τα πλαστικά των διαφορών χρωμάτων που, ε, για τα οποία γίνεται διαλογή, αλλά και για τα υπόλοιπα. Ε, να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε δηλαδή χωματερές ε, και κάποια από αυτά τα απορρίμματα δεν μπορούν να καούν, να καούν οπότε ε, θα πρέπει να ψάξουμε άλλες λύσεις και δεν μιλάω καν για τα ε, λάστιχα ας πούμε τα φθαρμένα εξαρτώμαστε κατά πολύ από τρίτε χώρε Πώς σκοπεύετε να λύσετε τέτοια ζητήματα στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ήρθε η ώρα για τις απαντήσεις και τα τελικά σχόλια. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Έλερ έθεσε πολύ σημαντικά θέματα. Το θέμα της, της βιομηχανίας της δημιουργικότητας. Ε, έχουμε τώρα ένα σύνολο εργαλείων για να υποστηρίξουμε την δημιουργική βιομηχανία, όπως ε, χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, το COSME, το INOFIN και η προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εσωτερική αγορά κτλ. Είχα μια ευκαιρία να συζητήσω με τους εκπροσώπους της Ιταλίας ε, πριν δύο εβδομάδες στον κλάδο της του κλάδου της δημιουργικότητας και ανέφεραν το θέμα των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ως πρώτο θέμα. Ανέμεναν μέτρα από την ευρωπαϊκή πλευρά. Το δεύτερο ήταν ότι η κυκλική οικονομία θα είναι μια κυριαρχή τάση και σε, πάρα πολλές, σε πάρα πολλούς τομείς της βιομηχανίας, της δημιουργίας. Μου είπαν ότι θα ήθελαν να είναι τμήμα των διαδικασιών της κυκλικής οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί θέλουν να μας βοηθήσουν να σχεδιάσουμε την πολιτική για να υποστηρίξει η πολιτική αυτή της ε, δημιουργικής βιομηχανίας. Πολλές από αυτές τις ε, κυρίαρχες ε, τάσεις ή τα οριζόντια εργαλεία πολιτικής που προτείνουμε αυτή τη στιγμή μπορούν να καλύψουν ε, μία σειρά τομέων ε, από τις ε, δημιουργικές βιομηχανίες μέχρι τις κατασκευές κτλ. Και αυτό μου οδηγεί στον οικολογικό σχεδιασμό, γιατί οδηγεί για τον οικολογικό σχεδιασμό. Είναι ένα καλό παράδειγμα για το πώς μπορούμε να δούμε τα πράγματα που θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της δημιουργικότητας, γιατί όσο πιο βιώσιμα είναι τα προϊόντα μας, τόσο υψηλότερο βρίσκονται στην ε, αλυσίδα αξία στην παγκόσμια αγορά. Και αν ε, μπορέσουμε να διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας αυτής, δυστυχώς δεν μπορώ να σας αναφέρω μια ημερομηνία, αλλά εξετάζουμε τις ε, δυνατότητες να διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογής όταν θα έχει οθετηθεί η νομοθεσία εδώ, αμέσως δημιουργείται ένα παγκόσμιο πρότυπο. Δηλαδή όλα τα προϊόντα που έρχονται στην ευρωπαϊκή αγορά θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια αυτά. Και ουσιαστικά σημαίνει ότι ε, προωθείται και η υψηλότερη ποιότητα που παράγεται από τους Ευρωπαίους. Κάτι άλλο που θα μπορούσαμε να κάνουμε, είμαστε ανοιχτοί σε καλές ιδέες γιατί ξέρω ότι ιδίω σε αυτό το τομέα χρειάζεται πρωτοτυποποίηση ε, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε υψηλή αξία και σε άλλους τομείς. Έτσι θα χρηματοδοτήσουμε την κοινωνία της πρόνοιας. Είμαστε όμως ανοιχτοί σαν έσυδες όπως σας είπα για το τι άλλο μπορούμε να κάνουμε, όμως πιθανότατα τα δύο μεγάλα θέματα είναι τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και η κυκλική οικονομία. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και ιδίως για το πρόγραμμα πλαίσιο 9. Κατανοείτε ότι δεν έχω όλες τις πληροφορίες που θα θέλατε να σας ε, αναφέρω. Θα προσθέσουμε την πρότασή μας στις 2 Μαΐου. Υπάρχουν ε, πολλοί κλάδοι που θα χάσουν χρήματα σε σχέση με το σημερινό πολίτες δημοσιονομικό πλαίσιο, όμως ε, υπάρχουν ε, κάποιοι τομείς όπου πιθανότητα θα δοθούν περισσότερα χρήματα και ο διάδοχος ε, του ορίζοντα 2020 θα λάβει περισσότερα κονδύλια και το Erasmus Plus είναι το δεύτερο πρόγραμμα που θα χρηματοδοτηθεί περισσότερο. Επομένως, πολλοί θα απογοητευτούν είτε επειδή θα χάσουν κάποια κονδύλια, είτε επειδή θα πάρουν τόσο όσα ήθελαν. Όμως αυτή είναι η πραγματικότητα λόγω του Brexit. Και είναι άλλη μια πραγματικότητα που πρέπει να λάβουμε υπόψη, γιατί πολλά κράτη-μέλη είναι κάθετα κατά της αύξησης ε, του μεριδίου του ΑΕΠ ε, για τον προπολογισμό της Ένωσης. γιατί δεν κατανοούν ότι έχει περισσότερο νόημα κάποια πράγματα να γίνονται μέσω του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού. Τώρα, το InFin και το Invest in EU. Ο στόχο μα είναι να δημιουργήσουμε ένα ταμείο Invest in EU που θα έχει τέσσερι θηρίδε πολιτική. Το ένα, η μία θηρίδα θα είναι για τι μικρέ και μισέ επιχειρήσει, το άλλο θα είναι η οι φόρες επενδύσεις, ε, μία άλλη θηρίδα θα είναι η κοινωνική και τώρα δεν θυμάμαι την τέταρτη. Όμως ο στόχος είναι να κατευθυνθεί η χρηματοδότηση στους τομείς πολιτικής που θα τεθούν ως προτεραιότητα από το Κοινοβούλιο και από τις Γενικές Διευθύνσεις. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχουν πολύπλοκα, ε, πολύπλοκοι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει λοιπόν να αντιγράψουμε το καλύτερο μοντέλο για την ναι. ενιαία κανονιστική πρόταση. Αυτό είναι σημαντικό και σε ό,τι αφορά το να κάνουμε περισσότερα με λιγότερα. Σύμφωνο ότι είναι ένα είδο δήλωση που χρησιμοποιείται ευρέω. Όμω το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων είναι ένα καλό παράδειγμα του πώς κάνουμε περισσότερα με λιγότερα. Αν δείτε το ποσό που επανακατανομήθηκε από διάφορες γραμμές προπολογισμών στο ΕΦΣΥ και αν το συγκρίνεται με αυτό που είχε το ΕΦΣΥ, τότε μπορούμε να πούμε ότι πράγματι κάνουμε περισσότερα με λιγότερα. Και η είναι δύναμη και πίσω από το Ταμείο InvestEU. Θέλουμε να ενεργοποιήσουμε το ιδιωτικό κεφάλαιο που είναι δυνατό και αν δεν είναι δυνατόν θα έχουμε επιχορηγήσεις. Τώρα, συμπληρωματι... το θέμα της ε, παρέκκλησης ε, της συμπληρωματικής προστασίας για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Θέλουμε να έχουμε ίσους κανόνες για τους παραγωγείς γενοσύμων σε σχέση με αυτούς που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτούς που βρίσκονται στις τρίτες χώρες. Δεν θέλουμε να θίξουμε ε, όλα τα SPC αυτά καθ' αυτά. Όμως το πρόβλημα σήμερα είναι όταν λήξει ο χρόνος προστασίας, οι ευρωπαϊκές εταιρείες δεν μπορούν να αρχίσουν να πουλούν αμέσω στις τρίτες χώρες. Κάτι που ισχύει με τις ευρωπαϊκές εταιρείε που έχουν έδρα σε τρίτες χώρες. Δεν ε, θέλουμε τώρα να αλλάξουμε καθόλου το πεδίο εφαρμογής ε, για το SPC, γιατί είναι ένα θεμελιώδες θέμα, αλλά θέλουμε να διατηρήσουμε ίσους κανόνες για τις εταιρείε ε, που έχουν έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με αυτές που έχουν έδρα σε τρίτες χώρες όταν θα έχει λήξει ο χρόνος προστασίας. Εδώ μιλάμε μόνο για τις ευκαιρίες εξαγωγής. Έτσι λοιπόν ελπίζουμε να έχουμε θετικό αντίκτυπο σε πολλά κρατημέλη και σε πολλούς κλάδους βιομηχανικούς. Ξέρατε ότι το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων έχει λειτουργήσει πολύ καλά σε διάφορες περιπτώσεις αποτυχίας της αγοράς. Αν δείτε τη χρηματοδότηση από το ΕΦΣΥ, κάθετο ΑΕΠ, η μεγαλύτερη πέντε είναι η Ελλάδα, η Εσθονία, η Βουλγαρία, η Πορτογαλία και η Ισπανία με τη σειρά αυτή. Έχουμε λοιπόν παροχή χρηματοδότησης ε, σε περιπτώσεις όπου δεν λειτουργεί επαρκώς η αγορά. Το ανανεωμένο ΕΕΦΣΥ υποτίθεται ότι θα παρέχει πολύ περισσότερα σε σχέση με το FC1 για την ε, αηφόρο επένδυση. Το 40% της χρηματοδότησης FC θα πρέπει να αφορά στόχους της ε, Συμφωνίας των Περισσίων για το κλίμα. Θα επικεντρωθούμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα λοιπά και φυσικά αυτό υποστηρίζει και άλλους στόχους πολιτικής μας. Τώρα, ποια πρέπει να είναι η κληρομιά αυτή τη Κομισιόν, θα πρέπει να κάνει η επόμενη Κομισιόν σε σχέση με τη βιομηχανική ανάπτυξη. Ανέφερα την κυκλική οικονομία. Πιστεύω ότι θα είναι το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα. Αν καταφέρουμε να έχουμε το κανονιστικό πλαίσιο. Η τεχνητή νοημοσύνη το δεύτερο, αν το χρησιμοποιήσουμε με έναν τρόπο που να βελτιώνει την ανάπτυξη και όχι μόνο την παραγωγικότητα, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη σίγουρα θα βελτιώσει την παραγωγικότητα, αλλά πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε και για την ανάπτυξη. Και το τρίτο στοιχείο είναι η ενδυνάμωση της ανθεκτικότητας ε, των ατόμων και των κοινωνιών σαν σύνολο. Τι εννοώ να επικεντρωθούμε σε εκπαίδευση ψηλότερου επίπεδου, γιατί θα πρέπει οι πολίτες μας να είναι ε, ικανοί να προσαρμοστούν, να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις. Δηλαδή δεν μιλάμε μόνο για την ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών, των κλάδων, αλλά και για την ανθεκτικότητα των κοινωνιών μας και των πολιτών. Γιατί αν χάσουμε τους πολίτες, ε, τότε δεν μπορεί η βιομηχανία να είναι ανταγωνιστική κυκλική οικονομία, τεχνητή νοημοσύνη και ανθεκτικότητα για τους ανθρώπους και μιλάμε κυρίως για την ποιότητα της εκπαίδευσης. Πολιτική ανταγωνισμού. Πολύ σημαντικό. Δεν είμαι ειδικό στον τομέα αυτό. Έχω ακούσει παρόμοιες απόψεις από πολλούς άλλους και δεν ξέρω αν κάνατε αυτή τη συζήτηση με την κυρία Στάκερ. Αν όχι, σας ενθαρρύνω να συζητήσω απευθεία μαζί τη γιατί μπορεί να σας δώσει πολύ καλύτερες απαντήσεις από μένα. Με συγχωρείτε. Λυπάμαι που σας διακόπτω. Δεν είναι καλή πρακτική και ζητώ συγγνώμη όμως δεν μπορείτε να απαντάτε αυτό. Είστε αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είστε ε, ένας πω αυτούς που είναι πιο κάθετοι στο να αλλάξουμε τους κανόνες ε, για την ε, κατάλληλη γεωγραφική αγορά. Δεν ξέρω γιατί λέτε ότι είμαι πάντοτε κατά της επαναξιολόγησης, γιατί ποτέ δεν έχω πει κάτι τέτοιο. Δεν θυμάμαι ποιο θα ήταν το πλαίσιο καν που να έχω πει κάτι τέτοιο. Όπως ξέρετε, υπάρχει ένα τύπος προστασίας μεταξύ της ε, ΓΔ και της υπόλοιπης ε, Κομισιόν. Δεν συμμετέχουμε στην ε, αξιολόγηση της αντίστοιχης αγοράς, αλλά έχω ακούσει παρόμοια παράπονα από άλλου, γιατί αλλάζει η αγορά. Κάτι που μπορεί να ισχύει σήμερα δεν ισχύει απαραίτητα αύριο. Γι' αυτό σας ενθαρρύνω να συζητήσετε με την κυρία Χέστινκερ απευθείας, γιατί ξέρετε τα πράγματα πολύ καλύτερα από μένα και αυτή η συζήτηση πρέπει να συνεχιστεί. Αυτή την άποψη έχω. Τώρα, φυσικά το θέμα το, του κόστου της ανταγωνιστικότητας πρέπει να λεφθεί υπόψη από τα κράτη-μέλη. Αλλά φυσικά ποτέ δεν θα μπορούμε να ξεπεράσουμε σε επιδόσει την ήπειρο τη φτηνότερη παραγωγή. Πρέπει να προστατεύσουμε του καταναλωτέ από τα φτηνότερα προϊόντα. Δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε εισαγωγέ από του άλλου. Όμω η καινοτομία και η προστάμενη αξία ε, μπαίνουν στην εξίσωση. Έχουμε, παραδείγματο χάρη, κάποιου γερανού που χρησιμοποιούμε στα λιμάνια μα. Έχουμε μια ευρωπαϊκή εταιρεία και μια κινέζικη εταιρεία. Και ένα ευρωπαϊκό λιμενέ αποφάσισε να ε, αγοράσει ένα γερανό που ήταν 25% ακριβότερο γιατί ήταν πολύ καλύτερη τεχνολογία και υπήρχε μεγαλύτερη ευφία. Υπήρχε μεγαλύτερη γνώση στους γερανούς αυτούς έτσι ώστε να αποφευθούν κάποια προβλήματα. Αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα ότι η τιμή δεν είναι το μόνο που μετράει. Λοιπόν, για το θέμα των πλαστικών. Πριν ε, δύο εβδομάδες παρουσιάσαμε τη στρατηγική για τα πλαστικά που σκοπεύει να δημιουργήσει μια καλύτερη νέα αγορά για τα απόβλητα πλαστικών. Θέλουμε να εναρμονίσουμε την ποιότητα των πλαστικών γιατί δεν μπορεί να λάβει χωρί ανακύκλωση σήμερα, γιατί έχουμε πάρα πολλές ε, ποιότητες ε, στα πλαστικά. Πολλές ιδιότητες. Αν σας ενδιαφέρει αυτό, σας συστήνω να εξετάσετε τη στρατηγική μας για τα πλαστικά, γιατί ε, έχει λάβει πάρα πολλές καλές κριτικές και από τη βιομηχανία, αλλά και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε πλαστικά, μια αγορά πλαστικών που θα βασίζεται στην κυκλική οικονομία και θα λειτουργεί καλά για να μειώσουμε τον όγκο των αποβλήτων και να χρησιμοποιούμε τα απόβλητα εδώ στην Ευρώπη και όχι να τα πουλάμε στις ασιατικές χώρες. Αυτό ήταν ένα πραγματικό πρόβλημα και γίνεται καθημερινά όλων και μεγαλύτερο πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ. Uh, thank Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αντιπρόεδρε, για όλες τις παρατηρήσεις σας, τις απαντήσεις που μας δώσατε. Σίγουρα ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που ακούσαμε και θα τα εξετάσουμε πολύ σοβαρά το θέμα, για παράδειγμα, του ανταγωνισμού γενικότερα. Ίσως η Επίτροφος Βεστάγκερ, που είναι αρμόδια για κάποια από τα θέματα αυτά, να μπορέσει να δώσει ικανοποιητική απάντηση στα ερωτήματά μας, διότι δεν είναι πρώτη φορά που προσπαθούμε να λύσουμε ένα τέτοιο πρόβλημα. Σας ευχαριστώ πολύ για όλες τις απαντήσεις σας. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη φορά. Uh, hello, once again, Madam Barbara Kappel. Βρίσκεται μαζί μας η κυρία Μπάρμπαρα Κάπελ, που είναι η συγγήτριά μας. Και έτσι περνάμε στο σημείο 6, επενδυτικά σχέδια σε ενεργειακή υποδομή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξέταση του σχεδίου έκθεσης. Στις 19 Δεκεμβρίου του 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της για κατάργηση του κανονισμού που απαιτούν από τα κράτη-μέλη να που βάλουν κοινοποίηση όσον αφορά έργα ενεργειακής υποδομής. Είναι η πρώτη φορά που εξετάζουμε το θέμα αυτό σύμφωνα με την κανονική νομοθετική διαδικασία. Κυρία ε, εισηγήτρια, έχετε το λόγο. Ε, σας ευχαριστώ κύριε ε, Πρόεδρε. Είναι πολύ σύντομο το σχέδιο έκθεσης αυτό. Χαίρομαι που μπορώ να παρουσιάσω ένα σχέδιο έκθεσης ε, που έχει να κάνει με το πλαίσιο REFIT. Πρόκειται για ε, κανονισμό που καταργεί έναν άλλον ε, κανονισμό, δηλαδή μείωση της γραφειοκρατίας και μείωση του άχθους. Θα ήθελα εκ των προτέρων να ευχαριστήσω τους κοιόδης εισηγητές για την καλή συνεργασία. Είχαμε πολύ θετικές συζητήσεις και σε επίπεδο βοηθών. Ε, χαίρομαι πολύ που υπάρχει γενική συμφωνία ότι θέλουμε καλύτερη νομοθεσία με το ε, πρόγραμμα REFIT. Ε, πολύ σύντομα να αναφερθώ στον κανονισμό. Μιλάμε για την κατάργηση ή πιθανή κατάργηση του κανονισμού που έχει να κάνει με την κοινοποίηση επενδύσεων σε ενεργειακές υποδομές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κανονισμός αυτός υιοθετήθηκε τον Φεβρουάριο 2014 ε, είχε να κάνει με την ε, πρόσβαση σε δεδομένα σχετικά με το δυναμικό και τα επενδυτικά σχέδια σε διάφορους ε, τομείς που έχουν σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και που έχουν ενδιαφέρον όσον αφορά την μελλοντική ενεργειακή πολιτική. Τρεις ε, φορές έχουν υποβάλει αναφορά τα κράτη-μέλη, το 2011, το 2013 και το 2014 και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατόπιν ε, στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΡΙΦΙΤ έχει αναθέσει τρεις εξωτερικές ε, έρευνες για να εξεταστεί η λειτουργία του κανονισμού αυτού. Το 2016 λοιπόν εκπονήθηκαν αυτές οι μελέτες, υπήρξε και δημόσια διαβούλευση που ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2016 και παρουσιάστηκε σε, σύντομη, ε, σε μια σύνοψη τον Νοέμβριο του 2016. Τα βασικά συμπεράσματα ήταν ότι υπάρχουν σημαντικές επικαλύψεις ανάμεσα στις ε, υποχρεώσεις κοινοποίησης του κανονισμού αυτού ε, και του, τις υποχρεώσεις σύμφωνα με το ENSO-E και το ENSO-G και επίσης οι περισσότερες πληροφορίες που διαβιβάστηκαν από τα κράτη-μέλη ε, ήταν πιο εύκολο να ε, αποκτηθούν μέσω άλλων ε, πηγών όπως είναι μέσω των δικτύων των διαχειριστών των δικτύων. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος της ε, για την παρακολούθηση της ενεργειακής αγοράς ε, διαθέτει σχετικές πληροφορίες. Έτσι λοιπόν θεωρήσαμε ότι μπορεί να ε, καταργηθεί ο κανονισμός για να μειωθεί το διοικητικό άχθος. Σύμφωνα λοιπόν και με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, πιστεύουμε ότι πρέπει να καταργηθεί ο κανονισμός 256 του 2014. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γιάμπορ, παρακαλώ έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ για την έκθεση αυτή. Επιτρέψτε μου να εκφράσω κάποιες αμφιβολίες σχετικά με την ε, πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την ε, έκθεση της εισηγήτριας. Ας πάμε λίγο πίσω. Ας εξετάσουμε την ιστορία της νομοθετικής αυτής πρότασης. Αρχικά η πρόταση της ε, Κομισιόν πήγε στο δικαστήριο, προσέφυγε το, το κοινοβούλιο, διότι θεώρησε ότι η νομική βάση ε, δεν ήταν η κατάλληλη. Η σύμβαση της Euratom δεν είναι το κατάλληλο, η κατάλληλη νομική βάση για ένα πρόγραμμα υποβολής κοινοποιήσεων. Κοινοβούλιο κέρδισε στην υπόθεση αυτή. Το δικαστήριο θεώρησε ότι θα πρέπει να έχει διαφορετική νομική βάση αυτός ο κανονισμός. Ποια ήταν η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της νίκης του Κοινοβουλίου, η κατάργηση του κανονισμού. Όχι να δεχτεί ότι θα πρέπει ο κανονισμός να υποβληθεί στην σωστή νομική βάση. Νομίζω ότι έτσι απλά παρακάμπτουμε το αποτέλεσμα της απόφασης του δικαστηρίου. Και δεν αποτελεί σωστή κατανόηση της απόφασης αυτής. Ε, τρία βασικά επιχειρήματα υπάρχουν από πλευράς της Επιτροπής για την κατάργηση του κανονισμού. Το πρώτο είναι η επικάλυψη όσον αφορά τις υποχρεώσεις κοινοποίησης. Και αναφέρθηκαν στα δίκτυα ένσω θεωρήθηκε ότι στο πλαίσιο των δικτύων αυτών ε, υποβάλλονται επαρκείς κοινοποίησεις. Ε, αλλά η υποχρέωση κοινοποίησης ε, σύμφωνα με έναν ευρωπαϊκό κανονισμό δεν μπορεί να αντικατασταθεί από υποχρέωση κοινοποίησης από πλευράς δικτύων όπου συχνά συμμετέχουν ιδιωτικές εταιρείες. Θεωρώ λοιπόν ότι οι υποχρεώσεις κοινοποίησης δεν αλληλοεπικαλύπτονται. Μπορούμε να σκεφτούμε πώς μπορούμε να ταιριάξουμε τα δύο αυτά μεταξύ τους. Δεν πιστεύω όμως ότι η κατάλληλη λύση είναι η κατάργηση του κανονισμού. Δεύτερο επιχείρημα. Έχουμε ήδη τρει κοινωνοποίησεις που υποβλήθηκαν, τρεις εκθέσεις υποβλήθηκαν. Ε, μόνο μία έχει υποβληθεί μετά το 2014 από τη θέση σε ισχύ δηλαδή του κανονισμού αυτού ε, και της εφαρμογής της Ενεργειακής Ένωσης. Ε, δεν πιστεύω λοιπόν ότι έχουμε επαρκή στοιχεία ε, μετά την ε, θέση σε ισχύ των ε, νέων κανόνων. Το άλλο θέμα που υπόθηκε είναι ότι υπάρχουν δυσκολίες όσον αφορά την εφαρμογή του κανονισμού στα κράτη-μέλη. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Εάν υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά την ε, εφαρμογή κανονισμού στα κράτη-μέλη, η απάντηση δεν είναι κατάργηση του κανονισμού αυτού, αλλά να ασκηθεί πίεση στα κράτη-μέλη ώστε να εφαρμόσουν καλύτερα τον κανονισμό αυτό. Και ε, συχνά αναφέρεται η καλύτερη νομοθεσία, αλλά και σε άλλα ε, τμήματα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας ε, η απάντηση είναι η καλύτερη νομοθεσία και όχι η κατάργηση της νομοθεσίας μόνο και μόνο επειδή υπάρχουν προβλήματα κατά την εφαρμογή της. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό που χρειαζόμαστε δεν είναι κατάργηση του κανονισμού και κλείνω κύριε Πρόεδρε. Η απάντηση λοιπόν δεν είναι ανάκληση, κατάργηση του κανονισμού αυτού αλλά να φροντίσουμε για την καλύτερη εφαρμογή του σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου και σύμφωνα με την ε, γραμμή του Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Αγαπητές συνάδελφε. Θα ήθελα τώρα να ζητήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την κυρία Εύα Γκέρχαρτς από την κυρία Διεύθυνση Ενέργειας για να σχολιάσει μιας και το θέμα είναι αρκετά σημαντικό για την Επιτροπή μας. Πείτε μας λοιπόν τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ναι, πρώτα απ' όλα η κυρία Γκερχάτ δεν είναι εδώ. Θα μιλήσω εγώ εκ μέρους της. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω αυτή την Επιτροπή για το σχέδιο έκθεσης που ε, αποδέχεται την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θυμίσω ποιοι είναι οι δύο βασικοί στόχοι αυτής της πρότασης. Καταρχήν να ξεφορτωθούμε με νομοθετική πράξη που δεν είναι πλέον χρήσιμη και δεύτερον να μειωθεί το διοικητικό άχθος για όλους τους εμπλεκόμενους στον κανονισμό. Τέλος, να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν το έκανε αυτό ε, ελαφρά την καρδία. Ε, ζητήσαμε πρώτα μια μελέτη από εξωτερικό συνεργάτη, ανεξάρτητη, για να δούμε τις τρεις διαδικασίες ε, ε αξιολόγηση το 2011, 2012 και 2013. Η μελέτη κάλυπτε και τις δύο ε, εκθέσεις, ε, όχι μόνο το 2011, το 2015, και είναι κάτι που συνοδεύει και τον κανονισμό περί διακυβέρνησης ε, του 2016. Θα θέλαμε να σα δώσουμε κάποιες σύντομε απαντήσεις στον κύριο Γιάβορ, αλλά και ακόμα ε, σε σχέση με κάποιε ανησυχίε που εξέφρασε. Πρώτα απ' όλα το θέμα της απόφασης. Ε, δεν καταργούμε τον κανονισμό λόγω της απόφασης. Αντικαθιστούμε τον κανονισμό βεβαίως που ακύρωσε ο κανονισμός, ο, το δικαστήριο, επειδή δεν αποφέρει τα αποτελέσματα τα οποία προσδοκούσαμε. Όχι λόγω της αποφάσης του δικαστηρίου. Και το δεύτερο στο οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Γιάβορ έχει να κάνει με τις δυσκολίες εφαρμογής του κανονισμού μέσω της ε, ε διαγραφής της κατάρριξης και όχι μέσω της βελτίωσης της εφαρμογής. Η αξιολόγηση που έγινε στη διάρκεια αυτών των τριών περίοδων μας έδωσε στο συμπέρασμα ότι τα προβλήματα στην εφαρμογή έχουν να κάνουν με τους περιορισμούς ε, τους δομικούς του κανονισμού. Μιλούμε εδώ για εκτιμόμενες δυνατότητες και αυτό ήταν κάτι το οποίο τα κράτη-μέλη δεν, μπορούσαν, δεν μπορούσαν να μας δώσουν ε, τουλάχιστον στο βαθμό ακρίβειας που ε, θέλαμε. Ήμασταν υπεραισιόδοξοι δηλαδή όταν ζητούσαμε ένα τέτοιο επίπεδο ε, πρόβλεψης, ακρίβειας πρόβλεψης. Και κάτι τελευταίο, ότι τώρα θα έχουμε δεδομένα μόνο από ιδιωτικούς φορείς. Το άρθρο 4 του κανονισμού που προτείνουμε να καταργηθεί ε, έλεγε ότι οι ιδιώτες θα δίνουν τις πληροφορίες στα κράτη-μέλη που στη συνέχεια θα αναφέρονται στην Κομισιόν τα δίνω αναφορά στην Κομισιόν. Και τώρα διαπιστώνουμε ότι η Κομισιόν ε, μπορεί να λάβει τις πληροφορίες αυτές άμεσα. και μέσω του δικού της παρατηρητηρίου που δίνει άμεση πρόσβαση ε, στις πληροφορίες από την αγορά χωρίς να περνάμε από διάφορους ε, ενδιάμεσους ε, ενώ τα στοιχεία ούτως ή άλλως από τις ιδιότητες προέρχονται τελικά. Αυτό Γι' αυτά είχα να πω. Να ευχαριστήσω την Επιτροπή για την πρόταση. Ευχαριστώ για τα σχόλια. Η εισηγήτρια τώρα. Τα τελευταία, τελευταία παρέμβαση. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Λεβόρ και ε, την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είχαμε τη δυνατότητα ε, να έχουμε ανταλλαγή απόψεων ε, και έχουν υποβληθεί και σχετικές ε, τροπολογίες. Οι προθεσμοί για την υποβολή τροπολογιών ε, είναι 26 του μήνα και ελπίζω μαζί να μπορέσουμε να πετύχουμε καλό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Μπάρμπαρα. 26 Απριλίου έως τις 12 το μεσημέρι την Πέμπτη, έτσι. Πέμπτη μεσημέρι η προθεσμία. Και ψηφοφορία στην Ήτρα 19 Ιουνίου. Το Σεπτέμβριο του 18 πιθανότατα στην Ολομέλεια. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας και για τις συζητήσεις που είχαμε. Αύριο το πρωί στις 9, 9 με 10 και κλεισμένο των θυρών μόνο συντονιστές στις 10 ψηφίζουμε. Να σας θυμίσω για άλλη μια φορά ότι ότι μία μισή με δυόμιση θα έχουμε την ολομέλεια ε, της κοινοβουλευτικής συνεργειακής κοινότητας. Ε, θα ήταν καλό να σας παραβρεθούν εκεί οι ευρωβουλευτές. Μία και μισή μεταξύ δηλαδή των δύο συνεδριάσεών μας της Επιτροπής Ήτρε. Θα έχετε και κάποιο σάντουιτς που θα σας περιμένουν εκεί. Σας περιμένουμε λοιπόν σε αυτή τη συνάντηση αύριο. Και βέβαια στις 10 αύριο το πρωί ψηφίζουμε στην Επιτροπή Ήτρε. Σας ευχαριστώ πολύ